Συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Είναι 3 και 5. Παρακαλώ μόνο μην κοιτάτε το ρολόι στα δεξιά, το αριστερό ρολόι να κοιτάτε, που πάει σωστά. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχω να κάνω μια ανακοίνωση το σημείο 19 αύριο ο Δανός Υπουργός Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης, ο κύριος Σον, ε, δεν θα μπορέσει να έρθει αύριο. Το σημείο 19 λοιπόν αφαιρείται από την ημερήσια διάταξη. Ε, θα ακούσουμε τον Δανό Υπουργό Μεταφορών αλλά ο Υπουργό Σον, ε, που είναι Υπουργό για την Αυτιλία, δεν θα μπορέσει να έρθει, οπότε αφαιρείται από την ημερήσια διάταξη. Είναι όλοι ικανοποιημένοι με την ε, ημερήσια διάταξη, με την τροποποίηση αυτή. Ωραία, εγκρίνεται. Δεύτερον, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 30 ε, και 31 Μαΐου. Ε, είσαστε όλοι ικανοποιημένοι με τα πρακτικά αυτά. Εάν ναι, εγκρίνονται. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα στη μεσαία διάταξη είναι η ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων. Πρόκειται για γνωμοδότηση προς την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ο κύριος Παγνιό, παρακαλώ. Euh, euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τις 15 Μαΐου, η ε, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η υποβόλη τροπολογιών, ε, συζήτησα με τον εισηγητή και τους όσους υπέβαλαν ε, τροπολογίες ε, ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς αύριο όσον αφορά το κείμενο. Οι τροπολογίες συμβιβασμού αφορούν τα εκτιμώντας 8 και 10. Η τροπολογία συμβιβαστική 2 καλύπτει τη ε, σημεία 18 έως 21 και λάμβανε υπόψη και τα υπόλοιπα σημεία που αφορούν την ηχοστάθμη των μηχανοκινητών οχημάτων, όπως η διευθέτηση των, των εδαφών και τα ελαστικά. Η τρο... συμβιβαστική τροπολογία 3 καλύπτει τις ε, τροπολογίες 26 και 27 και αφορά τις ελάχιστες ε, ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά και ευρεδικά αυτοκίνητα όσον αφορά τα παραρτήματα και ειδικότερα το παράρτημα 3 για τις οριακές τιμές. Ήταν πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό μεταξύ των μερών, των οποίων οι θέσεις ε, ήταν αντιδιαμετρικά αντίθετες. Παρ' όλα αυτά καταλήξαμε σε συμφωνία με τον σκιώδη εισηγητή, την κυρία Κοζά του ΕΛΚ, η οποία υπερασπιζόταν μια πιο ήπια θέση από τις υπόλοιπε ομάδες. Η συμβιβαστική τροπολογία 1 λοιπόν προτείνει μείωση της ηχοστάθμης κατά 4 δεσιμπέλ εντός 8 ετών, δηλαδή 2 δεσιμπέλ 2 χρόνια μετά από τη θέση ισχύ του κανονισμού, 2 δεσιμπέλ 6 χρόνια μετά και οριστικά 8 χρόνια μετά στο σύνολο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην αγορά, που στην αγορά. Ε, συμφωνούμε λοιπόν με τις τιμές που προτείνει η Κομισιόν, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ανησυχίες που διατυπώνει η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, παρατείνοντας την περίοδο προσαρμογής. Υπενθυμίζω λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι αύριο 9 το πρωί θα ψηφίσουμε ε, για το κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Πανιό. Ε, Ο κύριος Κόζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σιγητή για ε, το εγγραφό του. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε εκτενείς διαπραγματεύσεις, εξαιρετικά ωφέλιμες. Ήθελα να τονίσω ειδικότερα ότι εμείς οι σκιώδεις συζητητές υπήρξαμε ιδιαίτερα ανοιχτό μυαλό προς ιδέες των άλλων, ακούσαμε προσεκτικά ο στον τον άλλο και χάρη σε αυτό στα πιο αντικρώμενα σημεία καταφέραμε αρκετά ευέλικτα να επιτύχουμε συμφωνίε. Όσον αφορά το προηγούμενο κείμενο, πιστεύω ότι ο συμβιβασμός μας επιτρέπει να επιτύχουμε το στόχο μας όσον αφορά τις ε, εκπομπέ ε, θορύβου των αυτοκινήτων. Όσον αφορά του κατασκευάστες, πιστεύω ότι οι κατασκευαστές θα είναι ικανοποιημένοι με τις εδώ απαιτήσει. Και αυτό είναι ένας από τους σκοπούς μας. Συζητήσαμε πολύ για την πολιτική μεταφορών. Πολλά από το αρχικό κείμενο αφαιρέθηκαν ε, με το πνεύμα της πολιτικής μεταφορών μας Πιστεύω και ελπίζω ότι θα υποστηριχθούν όλες αυτές οι, όλοι αυτοί οι συμβιβασμοί. Πιστεύω ότι οι τροπολογίε βαίνουν προ την κατεύθυνση και ελπίζω ότι θα τη χάνουν υποστηρίξει. Um, ε, Ευχαριστώ, κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ, θα ήθελα να μιλήσω αγγλικά ε, διότι μιλώ εκ μέρους ε, του συζητή μας, που δεν μπο... της σκιώδους συζητήτριας, η οποία δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα και μου ε, έδωσε κάποιες σημειώσεις. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδους συζητητές για την καλή δουλειά που έχουν κάνει σε ένα πολύ τεχνικό θέμα. σε ένα θέμα που έχει υποβάλει σε εμά η Κομισιόν. Η ηχοσταθμή των μεταχυνήτων οχημάτων είναι σημαντικό θέμα, διότι ο θόρυβος αυτός επηρεάζει πολύ του ανθρώπου. Θα πρέπει να κάνουμε όσο γίνεται πιο πράσινε τις μεταφορές, αλλά θα πρέπει να να θέσουμε συγκεκριμένου ε, στόχους. Όσον αφορά τι ε, τροπολογίε, ε, μπορούμε να στηρίξουμε πολλέ από αυτέ, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία όπου δεν μπορούμε να στηρίξουμε τον εισηγητή. αυτό σχετίζεται με το παράρτημα 3, με τον πίνακα που βρίσκεται εκεί. Καταρχήν, η Κομισιόν δεν έχει συμπεριλάβει τον σχετικό τομέα όταν δεν άκουσε τις απόψεις ε, του σχετικού τομέα ε, κατά την προετοιμασία της πρότασης ή αν ακούστηκαν ε, σίγουρα δεν έχει λάβει υπόψη της τις θέσεις αυτές. Χρειάζονται σωστές αναλύσεις προτού να μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε τον πίνακα αυτών. Θα πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους. Ο κλάδος ε, μπορεί να μην θέλει να δαπανίσει τόσα χρήματα, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε την ε, ίδια κατάσταση ε, που είχαμε με τα όρια για το θιάφι στα καύσιμα για την αυτιλία, όπου δεν έγιναν διαβουλεύσεις με τον σχετικό τομέα. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί η Κομισιόν θέλει να διατηρήσει την κατηγοριοποίηση του 1985 για τα μηχανοκίνητα οχήματα, διότι έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε και έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Εγώ προτείνω η Επιτροπή να στηρίξει την τροπολογία μου υπαριθμός 70 ή να στηρίξουμε εμείς ε, την ε, τροπολογία 67 του κυρίου Κόχ και να καταψηφίσουμε τον πίνακα στο παράρτημα 3 και να ζητήσουμε από την Κομισιό να υποβάλει νέο ρεαλιστικό πίνακα λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση στην αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων. Ε, στην άλλη δεν αρέσει η συμβαστική τροπολογία 1. Εάν υπερψηφιστεί αυτή, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να καταψηφίσουμε το σύνολο της πρότασης ε, λόγω των όσων μόλις ε, σας διάβασα ε, που αφορούν τη θέση της κυρίας Σαβασάρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κράμερε για τους πράσινους. Μάικλ, παρακαλώ. Ο ε, σκιώδης εισηγητής μας, ο κύριος Κιστέλα, δεν είναι παρόν, ε, αλλά εκ μέρους του θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και τους σκιώδης εισηγητές. Θα είμαι πολύ σύντομος. Εάν οι συμβαστικές τροπολογίες οδηγήσουν σε αποδυνάμωση της πρότασης της Κομισιό, τότε θα την καταψηφίσουμε. Εάν ε, αποδυναμωθεί η πρόταση της Κομισιόν, ε, θα την καταψηφίσουμε. Αυτό είναι υπερβολικό για μας, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ευχαριστώ, κυρία Φώστερ. Τζάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή που οργάνωσε την ε, συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Δυστυχώ. μάλλον ε, να ξεκινήσω από τα θετικά. Όλοι θέλουμε να καταλήξουμε σε μια θετική λύση και θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται λιγότερη χορύπανση στου δρόμου μα σε όλον τον κόσμο, πόσο μάλλον στην Ευρώπη. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να το πετύχουμε αυτό με πρακτικά μέσα. Επικροτώ τις παρατηρήσεις της κυρίας Μάισνερ διότι είναι οι παρατηρήσεις που έκανα και εγώ εκ μέρους ε, της πολιτικής ομάδας ECR στην ε, συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Ε, θέσαμε ερωτήματα σχετικά με τα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει και στους, και στους τρόπους με τους οποίους γίνονται οι μετρήσεις. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες πληροφορίες. Καταλαβαίνουμε ότι έγινε μελέτη αντικτύπου, αλλά όταν πήρα το λόγο για το θέμα αυτό, την τελευταία φορά που ε, ανταλλάξαμε απόψεις. Ε, ρώτησα με ποιους ε, μηχανικούς μιλήσατε, μηχανολόγους, διότι εδώ δεν βλέπω να υπάρχουν κατασκευαστές μηχανών αυτοκινήτων και γι' αυτό ρωτώ πώς κατέληξαν στα νούμερα αυτά. Συμφωνώ με την κυρία Μάισνερ. Μήπως μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς καταλήξαν στα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα. Θα ήθελα πολύ να το γνωρίζω αυτό και νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι μας θα θέλανε. Ε, εγώ ανησυχώ και δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Ε, ακόμα και αν η Κομισιόν υποβάλλει σχετικό χρονοδιάγραμμα. Ε, εμείς κοιτάμε το, την αλυσίδα τροφοδοσίας ε, και τις εξαγωγές. Ε, τα στοιχεία αυτά αφορούν πολύ μεγάλο μέρος της αλυσίδας αυτής. Οι, οι μας ξέρω ότι κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να υποβάλουν τις τροπολογίες αυτές, αλλά λυπάμαι που η Κομισιόν δεν έχει απαντήσει σε μένα σχετικά με τα ερωτήματα που έθεσα και τις απαντήσεις που ήθελα σχετικά με το τι λένε οι μηχανολόγοι για αυτά. Και ε, ε, εάν καταλήξει κανείς να έχει μια πιο ήσυχη μηχανή, τι γίνεται με την κατανάλωση καυσίμων. Τέτοια ερωτήματα έθεσα και θα ήθελα πολλή απάντηση σε αυτά. Ε, με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας ε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε την πρόταση. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Αυτή είναι η θέση του, της πολιτικής ομάδας ECR αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Κομισιόν, παρακαλώ. Όχι. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μου δίνετε και πάλι ευκαιρία να σχολιάσω αυτό το θέμα ενώπιόν σας διαπιστώνω ότι παραμένουν ε, τα ίδια ερωτήματα όπως και την περασμένη φορά. Ορισμένοι θεωρούν ότι υπερβάλλουμε, άλλοι πάλι το αντίθετο. Απαντώντας την κυρία Φώστερ, σχετικά με το πώς καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα, λοιπόν είναι προϊόν συμβαστικής λύσης που εδράζεται σε μια ευρεία διαβούλευση επί σειρά ετών. Αυτή η νέα μέθοδος ε, δοκιμών ε, δοκιμάστηκε για τρία χρόνια για την πιστοποίηση των οχημάτων. Βασίσαμε λοιπόν την πρότασή μας στη βάση δεδομένων που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας. Αυτό το σχέδιο πρότασης ε, ως προς τη μέθοδο δοκιμής πάντοτε συζητήθηκε από, στη Γενέβη από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ ε, και χρησιμοποιούμε τα πορίσματα των εργασιών τους. Καταθέσαμε δε την πρόταση σε όλους τους ενδιαφερομένους. Συζητήθηκε επίσης στο ΚΑΡΣ 21 η πρόταση και γι' αυτό το λόγο καταθέτουμε όσο είχε την πρόταση στην Επιτροπή και υπενθυμίζω ότι συνιστά συμβαστική λύση που ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους. Ευχαριστώ. Κύριε Πανιό, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Δεν θέλω να ε, ρωτήσω κάτι. Αυτή η πρόταση που καταθέτουμε από κοινού με τον κύριο Κόζε, κυρίως ως προς το παράρτημα 3, ε, μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε ένα σημείο ισορροπίας. Είδατε από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων ότι υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων. Αφενός κάποιοι τα θέλουν όλα και τώρα για να μειώσουμε πολύ σημαντικά την ε, στάθμη του θορύβου μη λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αυτοκινητοβιομηχανία και από την άλλη πλευρά ε, υποστηρίζονται οι τροπολογίες που ικανοποιούν αυτή την ίδια αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτοί λοιπόν που θέλουν ε, τα πάντα δεν λαμβάνουν υπόψη την ε, μελλοντική βιομηχανική πολιτική. Κάποιος που έρχεται όπως εγώ από την Βόρεια Γαλλία επιδιώκει πάντοτε την εξέβρεση μαστικής λύσης. Ε, λοιπόν, για το παράρτημα 3, η λύση αυτή μας επιτρέπει να προχωρήσουμε, παραμένοντας όμως ε, ρεαλιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Φώστελ, διαδικαστικό. Ναι, επιτρέψτε μου ένα διαδικαστικό. Μάλλον ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγγνώμη, οι επιχειρήσεις δεν βασίζονται σε συμβαστικές λύσεις. Πρέπει να βασιζόμαστε σε δεδομένα, στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι να καλή είναι η πρόταση για την συμβαστική λύση. Πώς δεν μπορούμε να πουλήσουμε μια τέτοια λύση και η μεγαλύτερη ηρωνία είναι ότι όλοι υποστηρίζουμε τις καθαρές εισαγωγικά τεχνολογίες τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θέλουμε να έχουν 68 δεσιμπέλ και βλέπουμε το πίνακα και τα μηχανοκίνητα λέμε ότι πρέπει να πέσουν στα 69 δεσιμπέλ. Α με εξηγήσει κάποιο. Εμεί ρωτήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σαφήνεια αν έχει πληροφορίε σχετικά με το πώ οι κατασκευαστέ μπορούν να εφαρμόσουν την πρόταση. Απάντηση δεν λάβαμε, οπότε είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Ξέρουμε βεβαίω ότι ότι όλοι εργάστηκαν σκληρά, αλλά είναι η ανησυχητικά όλα αυτά. Εντάξει, θέλει η Επιτροπή να απαντήσει, μήπως το ερώτημα της κυρίας Φώστερ. Όχι, δεν νόμιζα και εγώ το θέλατε, οπότε θα δούμε. Θα δείξει αύριο στην ψηφοφορία θα δούμε τι θα κάτσει που λένε. Ε, τον Ιούλιο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εμείς αύριο θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πάμε στο επόμενο σημείο. Εξέταση τροπολογιών σχετικά με το e-call. Έχουμε την, τους δύο εισηγητές από τις Επιτροπές ΙΜΚΟ και ΤΡΑΝ. Θέλετε εσείς να αρχίσετε και μετά να ακούσουμε την εισηγήτρια από την ΙΜΚΟ. Με ποια σειρά θέλετε. Ο κύριος λέει κυρίες πρώτα. Παρακαλώ λοιπόν, σας ακούμε. Ε, Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Α, ε, ξαναπαίρνω τον λόγο, διότι όπως φαίνεται πρέπει να περιμένουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Μπορούμε λοιπόν, αν επιτρέπετε, να περιμένουμε πέντε λεπτά. Θα μπορούσε κάποιος να ψάξει να τον βρει, τον πρόεδρο της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Δυστυχώς πρωτόκολλο είναι, ζητώ συγγνώμη. Δεν είχα αντιληφθεί ότι έπρεπε να βρίσκεται εδώ. Okay, colleagues. Συνάδελφοι, ε, Όλγα πρώτη να μας ε, μιλήσει για την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Είμαι η συγγήτρια για την ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ συνάδελφοι, είναι η τρίτη συνεδρίαση μεταξύ Τραν και ΙΜΚΟ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή Ντίτρ Κοχ και όλους τους κοιόδης συζηγητές για την επικοδομητική και θετική του συνεργασία. Πιστεύω ότι έχουμε πλησιάσει ένα καλό τελικό αποτέλεσμα. Έτσι η εκθεσή μας θα στείλει ένα καθαρό μήνυμα υποστήριξης για την εισαγωγή του e εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Διεπιτροπών μας. Όπως ενημερώσαμε τους κοιόδης συζητητές μας την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, ο Ντίτερ και εγώ προετοιμάσαμε 31 συμβιβαστικές τροπολογίες που καλύπτουν όλα τα θέματα της αρχικής έκθεσης. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ξανά ευχαριστήσω όλους τους κοιόδη που έστειλαν τα σχόλιά τους μέχρι την περασμένη Παρασκευή. Προσπαθήσαμε να τα ενσωματώσουμε όλα και στην τελευταία στη λίστα τελευταίες ψηφοφορίες, ειδικότερα δύο σχόλια για την τροπολογία 14 όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που λάβαμε από το ΑΛΔΕ και το ECR. Την δεχθήκαμε με μια μικρή προσθήκη και ελπίζω ότι θα υποστηρίξετε αυτή, αυτό το συμβιβασμό. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τη συμβιβαστική τροπολογία 2 εμείς και οι Σκιώδης ε, συζητήσαμε κατά πόσο έπρεπε ή όχι να ονομάζουμε τις τρεις χώρες, να κατονομάζουμε τις τρεις χώρες που δεν υπέγραψαν το μνημόνιο συνεννόησης και συμφωνήσαμε με τον Τίτερ ότι πρώτα θα ψηφίσουμε τη συμβιβαστική χωρί τα ονόματα των τριών χωρών και μετά θα ψηφίσουμε ξεχωριστά το κατά πόσο θα κατονομάσουμε ή όχι αυτές τις τρεις χώρες. Και μετά ο κύριος Κοχ θα σα αναφέρει αργότερα περισσότερους συμβαστικέ και περισσότερα σχόλια. Ήθελα να πω ότι συνεργαστήκαμε εξαιρετικά καλά, βρήκαμε κοινή γραμμή από την αρχή με τους συνεισηγητές. Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο, δεν ήταν εύκολο, διότι προερχόμαστε από διαφορετικές ομάδες και διαφορετικές επιτροπές. Ωστόσο τα καταφέραμε. Αυτό αποτελεί ακόμη μια ένδειξη του πόσο θετική εικόνα έχει η ΙΜΚΟ ε, ως υπευθύνη για την οδική ασφάλεια. Επιθυμώ να στείλω ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αυτό αναμένει ένα μήνυμα από εμάς το οποίο θα αποτελέσει υπόδειγμα για τη νομοθετική πρόταση που ανακοινώνει για το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριο Κόχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα έλαβα μια γερμανική εφημερίδα όπου λέει ότι στην ε, οδό Α3 έγινε ατύχημα ε, στον αυτοκινητόδρομο ε, και δεν το πρόσεξε κανένας και Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να είχε υποφεληθεί από το e-call, από την ηλεκτρονική κλίση. Ε, θα ήθελα πάντως να ευχαριστήσω ε, όλους τους ε, συναδέλφους που έχουν ε, υποβάλει τροπολογίες. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε συμπεριλάβει όλες τις τροπολογίες, έχουμε βρει συμβιβασμούς, δεν έχουμε απορρίψει καμία τροπολογία. Δεν υπήρχαν άλλωστε σημαντικές ε, διαστάσεις απόψεων. να αναφερθώ σε κάποιες ε, συμβιβαστικές ε, τροπολογίες, την τέσσερα, όπου αναφερόμαστε στους στόχους και στα πιθανά ωφέλη. Βελτίωση της διαχείρισης των ατυχημάτων, μείωση των ε, ε, ε, σημείων συμφόρησης λόγω ατυχημάτων, θέματα ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση ατυχημάτων. Στην συμβαστική πρόταση 5 αναφερόμαστε στην αγορά εξοπλισμού. Δεν θέλουμε να πρέπει να υποχρεωτικά να εξοπλιστούν όλα τα παλαιά οχήματα με νέα συστήματα. στην συμβαστική τροπολογία 6 Έχουμε συνδυάσει διάφορες προτάσεις που έχουν υποβληθεί και καλούμε την Κομισιόν να σκεφτεί μήπως για τον γεωργικό τομέα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα για τρακτέρ και τέτοια. Τώρα αναφερόμαστε στα ε, ΙΧ και στα μικρά ΔΕΛΤΑΧΗ. Ε, αλλά βέβαια ε, ε, εισάγουμε και την πρόταση να ε, γίνει κάτι παρόμοιο με τα μεγάλα οχήματα, τα βαρέα οχήματα. Όσον αφορά την αναγνώριση των προτύπων, είναι και αυτό κάτι που μας απασχολεί. Έχουμε συζητήσει την δημόσια πρόσβαση στο σύστημα, το σύστημα δεν θα πρέπει όμως να είναι ανασφαλές. Πολλοί ε, συνάδελφοι φοβήθηκαν ότι θα δυσκολευτεί η πρόσβαση και γι' αυτό έχουμε διευκρινίσει καλύτερα την διατύπωση. Να υπάρχει πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και σε άλλους ε, ε, παρόχους υπηρεσιών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, διότι οι συμβαστικές τροπολογίες αντικατοπτρίζουν τις προτάσεις των συναδέρφων. Ε, άλλωστε έχουμε την ε, ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Η κυρία Γκούρμα ε, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, ΔΙΤΑ. ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν ε, πάντα χαίρομαι. Καταρχήν χαίρομαι που είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και όπως σας, είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση, Μα ενδιαφέρει η προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πρόσβαση στα συστήματα e-call παντού. Ήταν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Είχαμε τη δυνατότητα συνάντησης με όλους τους κοιόδες εισηγητές ε, στην αρχή. Και την προηγούμενη εβδομάδα, στην Σύνοδο του Στρασβούργου, Πιστεύω ότι μπορέσαμε να οροστικοποιήσουμε ε, τους συμβιβασμούς, ε, τις συμβαστικές προτάσεις που είναι πάρα πολύ καλές και μάλιστα η προθεσμία ήταν σήμερα το μεσημέρι. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν πολύ καλή η συνεργασία. Είναι πολύτιμη η ζωή κάθε ανθρώπου και γι' αυτό όλα τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στο e-call, όπως είναι και το δικό μου, θα πρέπει να σκεφτούν πόσο σημαντικό είναι το σύστημα αυτό. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι για την συνεργασία και ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι να μπορούν να έχουν τόσο ομαλές συνεργασίες. Και ε, ευχαριστώ και τον κύριο Κούσε για την ε, τροπολογία του διότι νομίζω ότι δίνει έτσι μια πτυχή ευαισθησία ε, ε, ε, στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Τίτα. Κάποιες συμβαστικές ακόμη δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Αυτό το τμήμα όπου κατονομάζουμε τους υπεύθυνου, θα πρέπει να το ψηφίσουμε ξεχωριστά. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει, διότι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν συμφωνήσαμε με αυτή τη συμβαστική τροπολογία είναι ακριβώς επειδή έχει αυτό το στοιχείο όπου καταλογίζουμε πράγματα σε κάποιους και ονοματίζουμε λόγος. Ε, name and shame. Σε σχέση τώρα με την 70... Δεν προσπαθούμε να κολλησιεργήσουμε, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται δοκιμή ε, και στα 27 κράτη-μέλη, όχι σε κάποια, πρωτού εφαρμοστεί στην πράξη, αλλά δεν νομίζουμε ότι αυτό συνεπάγεται μεγάλη καθυστέρηση. Πάντω ε, κάποιοι μας είπαν ότι προσπαθούμε να το θάψουμε κάτω από το χαλάκι και να καθυστερήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Δεν ε, συμβαίνει αυτό. Για την επέκταση των κατηγοριών για την ταξινόμηση, Χρειάζεται ανάλυση για, τα τρακτέρ, για τα ε, μηχανήματα εξκαφής. Ε, χρειαζόμαστε δοκιμές ε, και όταν μιλάμε για μηχανοκίνητα με τέσσερις ε, τροχούς, ε, όχι δύο. Επίσης χρειάζονται δοκιμές. Ε, δεν έχουμε καμία ένσταση για την επέκταση για να καλυφθούν και τα, όχι, τα φορτηγά. Ε, θα ακριθεί αυτό από τις υπόλοιπες ψηφοφορίες. Σχετικά με την τροπολογία της Νέτα για την προστασία των δεδομένων, Πρόκειται για την τροπολογία 14. Έχουν λυθεί τα προβλήματα που είχαμε. Thank you. Mrs. Ευχαριστώ. I'm sorry I came a little bit late. Uh. Συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά ήμουνα σε άλλη συνεδρίαση. Και πάντοτε συμβαίνει αυτό στο κοινοβούλιο. Έχουμε πέντε πράγματα να κάνουμε ταυτόχρονα κάθε φορά. Αυτά που βλέπω είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Όταν επεξεργαζόμαστε τόσο συγκεκριμένα θέματα, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια διακομματική συνεννόηση, ε, διότι το ύψιστο μέλημά μας είναι η ασφάλεια, λαμβάνοντας ε, υπόψη φυσικά και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Η επίτευξη αυτή τη ισορροπία ακριβώ ω προ αυτό το θέμα βρήκε μια πολύ συγκεκριμένη έκφανση και όπω είπε και η συγγήτρια και ο και ο συγγητή, δεν σημαίνει αυτό πρώτη φορά όπου ε, διακομματικά καταλήγουμε σε ικανοποιητικέ ε, συμβαστικές λύσεις. Εδώ ε, επιπροσθέτως έχουμε και δύο διαφορετικές συναρμόδιες επιτροπές ε, και τονίζουμε τα ουσιαστικά, δηλαδή ασφάλεια, ρεαλιστικές λύσεις και πραγματικά έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση που έχουμε αναχείρας, σε συμβαστικές τροπολογίες είναι μεν ουσιαστικέ, αλλά δεν θα έπρεπε να επικρατούν στη συζήτηση. Διότι στο μέλλον, αν καταφέρουμε να ε, καταθέσει νέα νομική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις λύσεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή ε, στην έκθεσή μας. Και ε, αυτό θα είναι ένα μεγάλο βήμα που θα έχουμε κάνει μετά από πολυάριθμα χρόνια ουσιαστικά άγωνων συζητήσεων. Έχει όντως συντελεστεί μια αλλαγή και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας. Ευχαριστούμε τώρα ο κύριος Τέλερ για... από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές, έκαναν εξαιρετική δουλειά με βάση τις δικές μου ιδεολογίες ή προτεραιότητες ε, που αφορούν το e-call ως μέτρο ασφαλείας, αφορούν την ελαχιστοποίηση των σοβαρών τραυματισμών, με την κινητοποίηση των υπηρεσιών εκτακτής ανάγκης ταχύτατα. Πιστεύω δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, γι' αυτό μας είπε ο κύριος Κοκ για το ατύχημα που δεν είχε ανακαλυφθεί για μερικές ώρες ε, και ήταν δύσκολο να εντοπιστεί, θα πρέπει να καταβάλουμε τις μεγαλύτερες δυνατές προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το σύστημα θα χρησιμοποιείται όσο πιο διαδεδομένα είναι δυνατόν. Όχι μόνο για τους οδηγούς και τους επιβάτες των αυτοκινήτων, αλλά για όλους τους χρήστες των οδών που ενδεχομένως εμπλέκονται σε ατυχήματα τα οποία κοινοποιούνται χάρη στον εξοπλισμό e-call. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την προστασία των δεδομένων, όπως αναφέρεται. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω δύο τροπολογίες δικές μου, 58 και 67. Η μία μιλάει για την αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής πιθανών εσφαλμένων συναγερμών μέσω της αυστηρών ελέγχων του συστήματος αυτού. Αυτό φυσικά είναι αυτονόητα και φυσικά παραμένει κάποια ασάφεια όσον αφορά το πώς θα χρηματοδοτηθεί η υποδομή. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να έχει διασαφενιστεί πριν ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τις οδούς τους. Θα πρέπει να μάθουμε δηλαδή ποιο θα τα πληρώσει όλα αυτά. Έχω συμφωνήσει με τις περισσότερες συμβαστικές και θα υποστηρίξουμε την τελευταία ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πόστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά ε, χαιρετίζουμε το εξαιρετικό σκληρό, τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει ο συγγητής και όλοι θέλουν σε αυτή την αίθουσα να καταλήξουν συμπεράσματα κατά πόσο μπορούμε να συμβάλλουμε στο να έχουμε τους πιο ασφαλείς δρόμους στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει διαφωνία στο ότι αν μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη υπηρεσία από τη σήμερα, τότε καλό θα έπρεπε να το κάνουμε με τη χρήση του αριθμού 112. Και φυσικά με ε, τη δυνατότητα των διαφορών φορέων, αστυνομία κτλ. να έρχονται σε επαφή με όλου. Αυτό δεν είναι καθόλου καλά, αλλά εδώ πιστεύω έχουμε ένα διτό ζήτημα. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι το ερώτημα κλειδί που θέτει ο κ. Στέιλορ. Μιλάμε για υποχρεωτικό εξοπλισμό με ένα τσίπι ενό κομματιού εξοπλισμού μέχρι το 2015 στα αυτοκίνητα και η ερώτησή μου είναι προς την Κομισιόν υπάρχει εγκαταστημένη όλη η υποδομή σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του τσίπ αυτού και ποιο είναι το προβλεπόμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας ε, το οποίο θα πρέπει να υπομισθούν τα κράτη-μέλη μαζί με όλες τις βελτιώσεις της υποδομές. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Όπως ε, ανέφερα λοιπόν ε, στις κάποιες τροπολογίες που υπέβαλα είναι ότι θα ήθελα να είναι εθελοντικό σύστημα εθελοντική δηλαδή η τοποθέτηση της συσκευή ε, σε ένα νέο αυτοκίνητο. Έχει υποβληθεί μια τροπολογία φυσικά που καλύπτει το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα και θεωρώ ότι αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να αξιολογούν και να αποφασίζουν μόνα τους, αλλά και το κόστος το οποίο έθεσα όταν το συζητήσαμε με την Κομισιόν για τους κατασκευαστές. Και εκεί υπάρχει μια διαφωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου παράγουμε περίπου 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα το χρόνο μιλάμε για κόστος 300 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ε, το κόστος υποδομών και το κόστος λειτουργίας. Δεν λάβαμε καμία απάντηση για όλα αυτά. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε αυτή τη στιγμή τι έχει να πει η Κομισιόν. Όπως ανέφερα υπάρχουν δύο ζητήματα. Ναι, από τη μια το υποστηρίζουμε ε, μετά ένα τρίτο μικρό ζήτημα ε, γενικού ενδιαφέροντος. Επειδή υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες, διαφορετικές υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος και φυσικά κάθε κυβέρνηση χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες και υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ε, εκτεκτής ανάγκης. Έχει μιλήσει με όλους αυτούς οι Κομισιόν, είναι έτοιμοι όλοι να προσυπογράψουν ένα τέτοιο σύστημα. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε εν ώψη των ψηφοφοριών τι έχει να μας πει η Κομισιόν Uh, Ο κύριος Χάρμπερ. Μάλκολμ, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για τη δουλειά που έχει γίνει πάνω στη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό παράδειγμα του πώς θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους οι επιτροπές, διότι όλοι επαφελούμαστε από τις προσπάθειες ε, του άλλου θα ήθελα να αναφερθώ στις πτυχές που ενδιαφέρουν περισσότερο τη δική μου επιτροπή και το πώς καταλήξαμε σε μια διαδικασία ε, με βάση και το δικό σας ενδιαφέρον για την, ασφάλεια, ε, για την οδική ασφάλεια. Το θέμα αυτό βασίζεται στην διαθεσιμότητα ενός ε, γενικού συστήματος ασφαλείας, το οποίο να μην περιορίζεται αποκλειστικά στο, στα αυτοκίνητα. Έχουμε ε, τον ε, πανευρωπαϊκό αριθμό 112, διότι υπάρχουν διαφορετικοί αριθμοί κλήσης στις διάφορες χώρες, στη χώρα μου είναι 999. και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι από το 2001 στην ε, ε, οδηγία για τις ε, οικουμενικές υπηρεσίες υπήρχε έκκληση προς τα κράτη-μέλη να κινηθούν προς ένα κοινό σύστημα στην κινητή τηλεφωνία και στα, ε, στις ε, επικαιροποιήσεις του 2008 και 2009 της πρότασης αυτής υπάρχει ε, απέτηση υπό την νομοθεσία τηλεπικοινωνιών προς όλα τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν τα δίχτυα κινητής τηλεφωνίας να μπορούν να επεξεργαστούν τα μηνύματα αυτά. Καταλαβαίνω αυτό που είπαν οι συνάδελφοι για το, για το κόστος, αλλά ε, το επιπλέον κόστος ε, για ε, το σύστημα αυτό σε σχέση με αυτό που ήδη έχουμε εδώ και 10 χρόνια είναι αρκετά χαμηλό. Εγώ έθεσα συγκεκριμένη ερώτηση προς την Επιτροπή την προηγούμενη φορά. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αλλά πρόκειται για μια, για ένα σημαντικό πρόσθετο μέτρο οδικής ασφάλειας που έχει, ε, που ε, βελτιώνει την ε, οδική ασφάλεια. Ο Ντίτερ Κόχ αναφέρθηκε στο σχετικό άρθρο. Δεύτερον, όσον αφορά τη δική μου εμπειρία, όσον αφορά την οδική ασφάλεια, πιστεύω ότι πράγματι έχει αποδειχθεί ότι το μέτρο αυτό σώζει ζωές. και στην κυρία Φώστερ ε, να πω ότι ε, με τον ίδιο τρόπο που δεν είναι προαιρετική η και δεν θα πρέπει να είναι ούτε και αυτό προαιρετικό. Τα περισσότερα κράτη-μέλη θέλουν ένα τέτοιο σύστημα και οι ε, κατασκευαστές θα θεωρήσουν πιο εύκολο να να έχουν σε κάθε όχημα το ίδιο σύστημα, κάτι που θα μειώσει και το κόστος. Σημαντικό θέμα που έχει τεθεί εδώ είναι ότι ήδη σε μεγάλο αριθμό οχημάτων ήδη υπάρχουν ιδιωτικά συστήματα ηλεκτρονικής κλήσης. Εδώ έχουμε ένα πρόσθετο βήμα. Και μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα αυτόματης εκκλήσης του αυτοκινήτου σε περίπτωση, για παράδειγμα, που γίνει ένα τύχημα και είναι ανέστητοι όλοι οι επιβάτες. γνωρίζουμε ότι σημαντικός αριθμός δεδομένων ε, συλλέγεται από τα σχετικά με ε, τον αριθμό των ατυχημάτων ε, και τη σοβαρότητά τους. Ε, συστήματα ηλεκτρονικών ε, αισθητήρων ε, αναπτύσσονται και θα εφαρμόζονται όλο ένα και περισσότερο. Θα είναι λοιπόν χρήσιμο τα κράτη-μέλη να επεξεργάζονται τα δεδομένα που να συλλέγονται με τα συστήματα αυτά. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω στην πρόταση αυτή. Τίνω να συμφωνήσω με τον κύριο Μενιάν. σχετικά με τη διεύρυνση του μέτρου αυτού ε, ώστε να καλύπτει και ε, βιομηχανικά οχήματα. Πιστεύω ότι θα είναι σημαντική αυτή η διεύρυνση. Από την άλλη όμως θα μπορούσαμε ε, να ενθαρρύνουμε τους κατασκευαστές ε, να το προσφέρουν ε, αυτό προς όλους τους πελάτες τους και έτσι να εισαχθεί πολύ πιο σύντομα το σύστημα αυτό. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα επιβατικά αυτοκίνητα και στην πλειοψηφία των ε, χρηστών των δρόμων. Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, πιστεύω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά. Πάντα μας ενδιαφέρει η προστασία των δεδομένων, ε, αλλά... Ε, βέβαια, τα θέματα αυτά αναφέρονται και στην οδηγία για τα δικαιώματα των χρηστών. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα πρότυπο το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από τα κράτη-μέλη σχετικά με τις εκκλήσει, που νομίζω ότι έχει μεταφερθεί με επιτυχία. Το δεν πρόκειται λοιπόν για νέα πτυχή, πρόκειται για κάτι το οποίο ήδη έχει καλυφθεί. Ε, γενικά Λοιπόν, πιστεύω ότι έχουμε μια σημαντική έκθεση η οποία ε, θα ε, ε, είναι καλό υλικό για την Κομισιόν και Στόχος είναι να ενσωματωθούν όλα αυτά ε, στον, ε, στο γενικότερο σύστημα 112 για όλη την Ευρώπη. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να αναπτυχθεί και το σύστημα εντοπισμού του, των, των κλήσεων. Υπάρχουν λοιπόν πολλά, συστήματα, πολλά, πολλές πτυχές τις οποίες μοιράζονται ε, τα δύο αυτά συστήματα. Ε, το πρώτο μνημόνιο κατανόησης ε, υπεγράφει το 2005-2006 για την ηλεκτρονική κλίση. Δεν πρόκειται λοιπόν για νέα ιδέα. Έχει έρθει όμως η ώρα να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μάρκο. Με δύο μιλητές έχω από την Κομισιόν, τον κύριο Ανίδια και τον κύριο Ζαν. Ο κύριος Ονίδη πρώτα. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά ξαναβρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας ε, και βλέπω ότι έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της ώστε να καλύπτει και πτυχή στη ΣΥΜΚΟ. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το κοινό έργο της δικής σας Επιτροπής και της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Επίσης είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τη δουλειά και των δύο συγκητών υπήρξε μια αρκετά έντονη ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιών για αυτό το σημαντικό θέμα. Το θέμα το οποίο μελετάμε εδώ και πολύ καιρό. Θέμα στο οποίο επίσης έχουμε επενδύσει αρκετές προσπάθειες και αρκετά χρήματα με πιλωτικά έργα και ούτω έκτιμα Εκτιμάμε ιδιαίτερα Αυτά που έχει, αυτό που έχει καθορίσει ο εισηγητής ως ε, σαφές μήνυμα το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο και σε ολόκληρη την Κομισιόν. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλές υπηρεσίε που ασχολούνται με το ζήτημα και να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να διατυπώσουμε μια εύλογη πρόταση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Για τις δαπάνες, θα έλεγα, για το κόστος, θα έλεγα ότι η τεχνολογία δεν είναι πρόβλημα. Ε, το κόστος, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς και μετά από τις συζητήσεις με τις διάφορες διευθύνσεις δεν είναι δυσβάσταχτο. Δεν είναι δυσβάσταχτο για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, ε, διότι η ευφυΐα χρησιμοποιείται παντού σήμερα στην τεχνολογία και έτσι η αυτοκινητοβιομηχανία μας έχει γίνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά. Το να προσθέσουμε λοιπόν αυτή την ειδική συσκευή που θα συνδέεται με το e-call δεν αποτελεί ουσιαστικά πρόβλημα. Αντιθέτως, ε, πρόκειται πιθανότητα για κάτι το οποίο θα βοηθήσει την ανάπτυξη μιας μεγάλης σειράς υπηρεσιών προστιθέμενης αξία. με ομαλό και αρμονικό τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και μετά από αυτό θα μπορέσει να επεκταθεί και παγκοσμίω. Δεύτερον, όσον αφορά την υποδομή, Πιστεύω ότι πολλοί από εσά μα υπενθύμησαν για τι υποχρεώσει που υπάρχουν δυνάμει τη τρέχουσα νομοθεσία. Και σε αυτή την ε, ε, περίπτωση ως υπεύθυνη της διατύπωσης των τεχνικών απαιτήσεων ε, για τις υπηρεσίες κλείσεων εκτάκτης ανάγκης μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το κόστος δεν αποτελεί ζήτημα το βασικό ζήτημα είναι οργανωτικό και υπάρχει και το ζήτημα εξέβρεση της σωστής διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων. Και σε αυτή την περίπτωση πιστεύω σε όλα τα κρατημέλη. Υπάρχει μεγάλη όρεξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή του e-call, διότι βάσει αυτού πολλές άλλες υπηρεσίες κρίσιμες για την οδική ασφάλεια, αλλά και για τις συνολικές τηλεματικές υπηρεσίες, μπορούν να αποτελεστούν δικημένο εκμετάλλευση, να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν σε ευρύτερη κλίμακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο συζητητές καθώς και τα μέλη των δύο συναρμοδίων επιτροπών για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους Κιώδης ε, για όλες τις ε, τροπολογίες. Λογικές φαίνονται οι συμβαστικές και η τελική διατύπωση μας βοηθά ώστε να συνεχίσουμε τις ε, σκληρές εργασίες των τελευταίων ετών ε, με στόχο την προώθηση των στόχων μας. Συμφωνώ με όλα αυτά που ακούστηκαν για το κόστος, αλλά ας μην ξεχνάμε και την εφέλη. Η αξιολόγηση αντικτύπου προβλέπει μεγαλύτερα ωφέλη από το κόστος που συνεπάγεται αυτή η δρέση. Λόγω οικονομία κλίμακα μπορούμε με μικρό κόστο να συμπεριλάβουμε αυτή τη δυνατότητα κλίση όλα τα οχήματα, αλλά όχι μόνο. Μπορούμε να καλύψουμε και τις υποδομές. Είπατε για την υπηρεσία εντοπισμού του καλούντος. Αυτό συνεπάγεται υποδομή, νέα υποδομή. με μία ελάχιστη προσάυξηση ως προς το αρχικά προβλεπόμενο κόστος για την ε, προαιρετική αυτή προσέγγιση. Το προσπαθήσαμε πολύ καιρό, αλλά δεν καταλήξαμε και γι' αυτό εξετάζουμε και άλλα εναλλακτικά σενάρια. Αυτά τα τρία σενάρια έχουμε υπολογίσει να λειτουργούν ταυτόχρονα, διότι θέλουμε οι υπηρεσίε να αρχίσουν να εφαρμόζονται ταυτόχρονα. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε και το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τις αρχές καθώς και με τον επόπτη των δεδομένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση Τώρα ως προς τις κατηγορίες των οχημάτων είναι ξεκάθαρο για τον, ε, τον αριθμό ενεργοποίησης για τα βαριά οχήματα. Υπάρχουν πάντως ομάδες εργασίας που συνεχίζουν να εξετάζουν αυτά τα θέματα στο Συμβούλιο και ίσως ε, θα ήταν πρόωρο να καλύψουμε όλες αυτές τις κατηγορίες ε, των οχημάτων αυτή τη στιγμή. Θα εξακριβώσω κάποια από τα στοιχεία για τα οποία με ρωτήσατε τις παρεμβάσεις και θα επανέλθω. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Ε, θέλετε να κάνετε τη συντομότερη δυνατή ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάμε για οχήματα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη και μιλάμε για την περίοδο μέχρι το 2015. Ωραία, αν αγοράσω εγώ ένα όχημα που έχει κατασκευαστεί σε τρίτη χώρα, ε, τι γίνεται τότε με τη συμπερίληψη αυτού του ε, εξοπλισμού που είναι υποχρεωτικός για όλα τα οχήματα που κατασκευάζονται εδώ στην Ευρώπη. Ποιος θέλει να απαντήσει. Malcolm, you answer it. Why they have a conflag, you answer it. Malcolm, ε, ε, είσαι, συγγνώμη, αρμόδιος, θα απαντήσεις. Ε. Αυτό λοιπόν, αυτός ο περιορισμός απάντηση ισχύει για όλα τα οχήματα που κατασκευάζονται εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εγκριθούν. Ούτως ή άλλως δεν μπορούν να απολυθούν αυτά τα οχήματα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες αν δεν συμπεριλαμβάνουν αυτό τον εξοπλισμό. Αυτό θα προβλεφθεί, θα το εξετάσουμε αυτό από κοινού με τους κατασκευαστές για να δούμε αν είναι διαθέσιμη η τεχνολογία. Ο κύριος Χάρμπορ, λέει ο κύριος Σίμψον, σίγουρα ξέρει για τι πράγμα μιλάει, αλλά θα ακούσουμε και την, ε, την Επιτροπή. Α, ναι, και προσθέτει ο κύριος Χάρμπορ ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα νέα και στα παλιά οχήματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, στη συνέχεια θα προκύψει. Ωραία, ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, και αύριο θα ψηφίσουμε. και τον Ιούλιο θα περάσει από την Ολομέλεια. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και εσείς Πρόεδρε της ΣΥΜΚΟ και τα μέλη της Επιτροπής. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε για αυτό το θέμα. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο σημείο. Πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014 2014-2020 παρουσίαση σχέδιο. <laughs> έκθεση, της δικιάς μου έκθεσης.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 Λοιπόν, εδώ ασχολούμαστε με την ενδιάμεση έκθεση ε, τη Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών για τι Προϊόντες Διαπραγματεύσει για το Πολιετέ Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το που όπω είναι οικείο σε όλου μα, ε, και βάσει των κανόνων ένα σχέδιο έκθεση ε, δεν μπορεί, εφόσον πρόκειται για μη νομοθετικού χαρακτήρα έκθεση και υποβάλλεται για μετάφραση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία σελίδα. Δεν γινόταν όμως να καλύψουμε όλα τα ζητήματα που ενδέχεται να ακύψουν μέσα σε αυτό το σχέδιο είναι πιθανό ότι θα κατατεθούν ε, πολυάριθμες τροπολογίες για το σχέδιο εκθεσίμου για να καλύψουμε ζητήματα όπως τα ταμεία συνοχής, ε, διαρθρωτικά ταμεία, θαλάσσια πολιτική, γκαλιλαίο κτλ. κτλ. Γι' αυτό εγώ προσπαθώ να τροποποιήσω τη δική μου την έκθεση γιατί μια σελιδούλα μόνο μας επιτρέπουν να έχουμε οπότε δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα σημεία. Είχαμε και μια πολύ μεγάλη έκθεση για το ψήφισμα τη Σούρε, αλλά εγώ επέλεξα διαφορετικό δρόμο. Ήθελα να είμαι σαφή, συνοπτικό και να ασχοληθώ με τα βασικά ζητήματα και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ακούσουμε τους κύριο Μπό και Κάλφιν, του συζητητέ από την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών και βεβαίω έχουμε την διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου για τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο που πρέπει να ακούσουμε 10 Ιουλίου είναι η προτινόμενη καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών, όμω δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων ε, επιδανικής προεδρίας ε, στι 18 8 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή. Οπότε και μετά το καλοκαίρι έχουμε χρόνο, έχετε χρόνο μόνο για να καταθέσετε τροπολογίες. θέλημένα έγινε αυτό. Ούτω ώστε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και σε άλλες επιτροπές, στο Συμβούλιο ούτω ώστε η Επιτροπή Μεταφορών να καταθέσει εν τέλει μία συνεκτική πρόταση. Υπάρχουν και άλλε πολύ ανησυχητικέ φήμες από πλευρά του Συμβουλίου. Φαίνεται ότι πολλά κάποια κράτη-μέλη και ξέρω ότι δεν μπορούμε εδώ στην Ένωση να κατονομάζουμε κάποιους, αλλά θα το πω. Η Γερμανία θέλει να περικόψει με πάνω από 50% το χρηματοδοτικό μέσο Connecting Europe. Η αντίδρασή μας ποια πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου, για την αναβάθμιση των υποδομών και για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπετε μέσα στο πρόγραμμα ΣΕΦ, ε, βάσει του ορίζοντα 2020, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε τη σημασία των μέσων για την ανάπτυξη και να αναγνωρίσουμε και το βάρος αυτών των τομέων της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξυπηρετούν άμεσα τη στρατηγική 2020. Στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου επίσης χρειάζεται δουλειά για να ξεκαθαρίσουμε ότι οι επενδύσει στον τομέα των μεταφορών έχουν στρατηγική σημασία, ούτω ώστε να μπορέσουμε να υπερβούμε την τρέχουσα οικονομική κρίση. Δράτω με τι ευκαιρίες λοιπόν, καλώ τους δύο εισηγητές για το πού Πουδουπού στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών, ούτως ώστε να τονίσουμε ε, το περιεχόμενο αυτού του σημαντικού μηνύματος. Ε, τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 31,3 δις ε, για 10 προγράμματα ε, που ε, θα υλοποιηθούν από τον αρμόδιο οργανισμό. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 8 δις που διαχειριζόμαστε με κεντρικό τρόπο υπό το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2013 δηλαδή τμήματα του ορίζοντα 2020 και συγκεκριμένα για τις ε, ευφυείς ε, πράσινες μεταφορές ε, καθώς και η εξασφάλιση της καθαρής και αποτελεσματικής τεχνολογίας. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο στο συνολικό ποσό των 6,3 δις ε, πιο υποτμήμα ε, ή μάλλον το υποτμήμα για τα καύσιμα δεν είναι ξεκάθαρο ποιο κονδύλι θα έχει. Ως προς την έρευνα είναι σημαντικό να παρα... διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ε, ρόλο στο τομέα της ε, βιομηχανίας ε, και πιστεύω ότι η έρευνα χρειάζεται και όλα τα τέντη προγράμματα θα υποφεληθούν από αυτή τη δράση. Τώρα για το Ταμείο Συνοχής θα έχει 34 δις χοντρικά για προγράμματα που σχετίζονται με τις μεταφορές και τα 10 δις για το ΣΕΦ, το Connecting Europe. Πρόκειται για μια βασική πηγή χρηματοδότησης για τις υποδομές μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν γέννη στηρίζουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίζεται στο τωρινό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά θέλω να αυξήσουμε τα ποσά που διαχειριζόμαστε κεντρικά, κυρίως στο χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, διότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να έχουμε τα ελάχιστα κονδύλια που χρειαζόμαστε. Θα ε, ε, προκρίνουμε επιπροσθέτως 10 δις ε, για το ΣΕΦ. Θέλουμε το ΣΕΦ να αναλάβει τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Επίσης θέλω να τονίσω την σύνδεση ανάμεσα σε κάποια προσδιορισμένα εκ των προτέρων προγράμματα, δηλαδή ε, στο παράρτημα του σχετικού κανονισμού και να τα συνδυάσουμε με τις προτάσεις που γίνονται για το ΣΕΦΕ στο επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε 31 θέσει που μπορούν να υποστηρίξουν τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών ο στόχος του Συμβουλίου είναι να έχουμε εθνικά ευχολόγια, χωρίς όμως να προσφέρουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι πρέπει να απορριφθεί αυτή η θέση. Αν θέλει το Συμβούλιο να μειώσει τα ποσά για το ΣΕΦ, πρέπει να μας πει ποια προγράμματα λοιπόν θα διαγραφούν από το συγκεκριμένο παράρτημα. Αναφέρθηκα επίσης ε, στην ανάγκη της συνέχισης του προγράμματος Μαρκοπόλο που αναμένεται να εκπνεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαίνεται ότι δεν επιθυμεί τη διατήρηση του προγράμματος ε, και θέλει να το βάλει στις κατευθυντήριες γραμμές ε, για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Το τωρινό πρόγραμμα έχει 450 εκατομμύρια στην τωρινή δημοσιονομική περίοδο και έχω την εντύπωση ότι τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν στο νέο ΣΕΦ για τη συνέχιση του προγράμματος Μάρκο Πόλο και γι' αυτό σας λέω ότι υποστηρίζω τη διατήρηση ε, του προγράμματος Μάρκο Πόλου ε, ως έχει. Αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία της πρότασής μου και όπως σας είπα και προηγουμένως Ε, προτιμώ να εξετάσουμε ένα μακρύτερο κατάλογο τροπολογιών και να αφήσουμε την ψηφοφορία για το Σεπτέμβριο, ούτω ώστε να μπορέσουμε με του σκιώδει να δηλώσουμε με σαφήνεια τι προθέσει τη Επιτροπή ε, Μεταφορών, ούτω ώστε να διαβαστεί το έγγραφό μα στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών και ευελπιστούμε ότι θα συμπεριληφθεί σε μια κρατέα θέση του Κοινοβουλίου που θα προβληθεί κατά τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου πιστεύουν ότι αν το Συμβούλιο επιθυμεί να περικόψει το ΣΕΦ θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς θα περικόψει. Ωραία, ευχαριστούμε. Γκράς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, στις διάφορες ομάδες εργασίας έχει συζητηθεί επανειλημμένα το θέμα αυτό και είναι σαφές ε, για μας ότι ο παρόν δημοσιονομικός σχεδιασμός ε, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ε, στην διευκόλυνση αυτή ότι ε, οι μεταφορές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του. Ελπίζουμε κάποια μέρα να μπορέσουμε να πείσουμε το Συμβούλιο να καταλάβει ότι ε, οι μεταφορές, ότι οι επενδύσεις μεταφορές είναι τριπλές. Καταρχήν όταν γίνεται η επένδυση αποτελεί ε, οι, οι επενδύσεις και άμεσα και έμεσα και μακροπρόθεσμα δηλαδή ε, ωφελούν ε, τις περιφέρειες και γι' αυτό Ελπίζουμε στη χρηματοδότηση από την Κομισιόν, διότι πιστεύουμε ότι Ε, αλλιώς ε, δεν θα μπορέσουμε να χτίσουμε ε, σωστά δίκτυα. Ε, στην Ευρώπη το θέμα λοιπόν είναι ο, όχι απαραίτητα να μειωθούν τα χρήματα για τα διάφορα προγράμματα, αλλά να, μειωθού, να μειωθεί ο αριθμός των προγραμμάτων ή των έργων αυτών. Θα θέλαμε ήδη τώρα να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα, διότι... θα πρέπει οι χώρες συνοχής να λάβουν απάντηση σε κάποια από τα ερωτήματά τους. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, χώρες ε, που γρήγορα μπορούν ε, να βρουν πόρους. Θα πρέπει να απαντήσουμε στα ερωτήματα των χωρών συνοχής. Και επίσης ε, το αν τα χρήματα βρίσκονται εντό του 2,5% ή εκτός ε, και αυτό θα πρέπει να το απαντήσουμε, θα πρέπει να υπάρχει ε, να δοθούν σωστές απαντήσεις επιπλέον. Γενικά, στις ε, μακροπρόθεσμες αυτές προοπτικές θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε τα μέσα αυτά που προβλέπονται εδώ. Ε, αν θέλουμε να πετύχουμε έστω και κατά το ίμιση τους ε, στόχους μας. Πρόκειται για ένα ελάχιστο ποσό αυτό που προτείνεται αυτό εδώ. Πιστεύω ότι παραμένει σημαντικό να έχουμε συνοχή ανάμεσα στις ε, εκθέσεις μας ε, για, το, για τη διευκόλυνση αυτή και ε, στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Επιπλέον θα ήθελα να θέσω το ερώτημα σχετικά με, τις, με τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό, διότι η διευκόλυνση αυτή αποτελεί ένα πυρηνικό σημείο για το μέλλον. Έχουμε και άλλους ε, τομείς. Ε, η έρευνα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχει ενισχυμένη θέση στον τομέα των μεταφορών. Ε, επικροτώ ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να εξετάσουμε την έκθεση αυτή, ώστε να μπορέσουμε μαζί να εκπονήσουμε ε, μία έκθεση η οποία να υποστηριχθεί από, την, ε, από ευρία πλειοψηφία στην Επιτροπή μας. Επίσης, ε, αν κοιτάξουμε την απορρόφηση των πόρων ε, στο τελευταίο διάστημα. Ε, πιστεύω ότι θα μπορέσει να αποτελέσει προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή πολιτική, ε, να στηρίξουμε έργα τα οποία μακροπρόθεσμα να επιφέρουν προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Γίνεται μια κατά τη γνώμη μου παράλογη συζήτηση ε, σχετικά με το ποια επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τα χρήματα. Το θέμα είναι να ε, ε, χρησιμοποιηθούν με τρόπο συνεκτικό τα χρήματα και προ όφελο όλων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καθότι ο σε ήδη είπε πολλά και ο Ματιό Εγκρό αναφέρθηκε σε αυτά, δεν χρειάζεται εγώ να πω πάρα πολλά. Ε, συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά ε, τον ε, προϋπολογισμό, τα, το, το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο κλπ. Η διευκόλυνση ε, για την Ένωση της Ευρώπης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, αλλά το κράτος μέλος από το οποίο προέρχομαι εγώ θέλει να μειώσει το ποσό αυτό και ε, ε, εξεπλάγει, διότι είδα τον χάρτη των διευρωπαϊκών δικτύων ε, και στην Βόρεια Γερμανία, για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνονται και τα εσωτερικά ύδατα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ενώ η Γερμανία ήθελε να αποκλειστούν. Εδώ έχουμε μια δυνατότητα όχι μόνο να προωθήσουμε την ενιαία αγορά και τις μεταφορές, ε, αλλά να ε, επανέλθουν ε, οι πόροι με λογικό τρόπο στις περιφέρειες. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντική η πρόταση αυτή. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το θέμα, ξέρω ότι θα πρέπει να πείσουμε σε πολλά επίπεδα ότι είναι καλή η πρόταση αυτή και θα είναι σημαντική για το μέλλον. Σημαντικό για μένα είναι να συμπεριλάβουμε και τα πιλωτικά προγράμματα. Ξέρω ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στο διάστημα 2014 με 2020, είναι από τώρα μέχρι το τέλος του 2013, αλλά θα είναι σημαντικά αυτά για την μελλοντική φάση. Κατά τη γνώμη μου είναι λογικό τα κράτη-μέλη να υπερασπίζονται περισσότερα την πρόταση αυτή της ε, Κομισιόν. Και έτσι ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε το χρηματικό ποσό που χρειαζόμαστε, διότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα από αυτά που προτείνονται. Ε, όσον αφορά την ε, συνοχή, αναφέρθηκε σε αυτό ο Ματιό, υπάρχουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ αυτά που θεωρούν τα κράτη ότι ότι τα χάνουν, αλλά ε, δεν ισχύει αυτό. Μήπως ε, θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα στα κράτη, ε, να αποφασίζουν δηλαδή, τα κράτη για μεγαλύτερο ποσό. Και επίσης, αναφέρθηκα ήδη στα εσωτερικά ύδατα, σημαντική για μένα είναι και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ε, και το χρειαζόμαστε αυτό για την βελτίωση της ενίας αγοράς. Ε, γενικά νομίζω ότι η γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής μας θα είναι συνενετική και πιστεύω ότι είναι καλό το ότι θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κράμερ εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για την παρουσίαση του θέματος. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια θέματα. Η νέα πολωνική κυβέρνηση ε, έχει απορρίψει την πρόταση της προηγούμενης κυβέρνησης. Είπαν ότι ε, τα τρένα υψηλής ταχύτητας ε, είναι θέμα για την Πολωνία σε 30 χρόνια και προσπάθησαν να εξηγιάνουν τον προϋπολογισμό και και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό, αλλά αν θέλουμε περισσότερα χρήματα χρειαζόμαστε ε, διαφορετική πολιτική ώστε να πετύχουμε περισσότερα ε, με τα χρήματά μας. Αν θεωρήσουμε ότι θα λάβουμε 10 ε, δισεκατομμύρια περισσότερο και ότι το τούνελ πρέπει να θα ολοκληρωθεί πιο γρήγορα, σε 30 χρόνια πάλι δεν κερδίζουμε τίποτα. Σημαντικό είναι να βάλουμε φρένο ώστε να αποφύγουμε τα χρήματα να πηγαίνουν αποκλειστικά στον τομέα των οικοδομών και όχι για να βελτιώσουμε τις μεταφορές. Επίσης, ε, στο γερμανικό Bundestag έγινε μια εσωτερική συζήτηση όπου ο καθηγητής Χέχτα από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου είπε ότι 20 με 30% ε, της ε, ε, ενέργειας μπορεί να εξοικονομηθεί με αυτόματα φρένα. Πολλές εταιρείες ε, μεταφορών όμως ήταν ε, κατά αυτού διότι ε, είπαν ότι τότε θα πρέπει να αλλάζουν πιο συχνά τα λάστιχα. Αλλά ένα τέτοιο αυτόματο φρένο τίθεται σε ισχύ μόνο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και μάλιστα μπορούν να μειωθούν και τα decibel. Ε, η ηχοστάθμη δηλαδή. Και αυτή θα ήταν μια θετική επένδυση. Θετικό βρίσκω επίσης ε, το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο. Μπράιαν αναφέρθηκε σε αυτό. Σε αυτό ξέρουμε ότι υπάρχουν προθέσεις ε, να καταργηθεί αυτό, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Σύμφωνα με τον κύριο Βαντάλεν, η αρχική σας δήλωση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ήθελα να πω ότι συμφωνώ με όσα είπατε κυρίω όσον αφορά το Europe Connecting Facility στα σημεία Ήθελα απλά να πω ένα επιχείρημα. Ορισμένα κρατημέλη θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μείωση του προπολογισμού για το, στο μισό του Connecting Europe. Εάν ταυτόχρονα απαιτούν ε, πολιτική ένωση, δημοσιονομική, οικονομική ένωση, πρέπει να καταλάβουν ότι όλες οι διαφορές ε, που υπάρχουν σε μια τέτοια πολιτική ένωση απαιτούν περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους. Συνεπώς πρέπει να σκεφτούμε, να λάβουμε υπόψη τα άλλα κράτη-μέλη και τις περιφερειακές ε, τις περιφέρειες της Ευρώπης. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την επιχειρηματολογία. Για ποιο λόγο πρέπει να μειώσουμε για την επόμενα δημοσιονομική προοπτική το Connecting Europe Facility κατά το μισό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που θέλουμε να δούμε στο μέλλον για το 2020. Θέλουμε μια ένωση με πολύ χαμηλό επίπεδο περιφερειών χωρίς σύνδεση με τα κεντρικά και τα δυτικά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα Εντελικά. τελικά. Ε, ευχαριστώ Πίτερ Βαντάλεν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας ε, δίνετε, μας προσθέσετε αυτό το πολύ καθαρό μήνυμα με αυτή την ε, πρόταση νομοδότησης. Ε, έχω μερικές ερωτήσεις. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδείξει την αξία του. Για την επιτυχία του προγράμματος αυτού ελπίζω να λάβετε υπόψη τις τροπολογίες μου στη παράγραφο που αφορά τις επενδύσεις στις υποδομές TNT, παράγραφος 4, έχω μια ερώτηση για την Κομισιόν. Αναφέρατε ότι θα υπάρξουν κάποιες περικοπές, γι' αυτό τι θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν ή το Συμβούλιο. Τι γίνεται με την υποδομή, με τη χρηματοδότηση των υποδομών. Τι γίνεται με αυτό το νέο κανάλι Northwood ε, που μπορεί να διακοπεί. Θα ήθελα να μας δώσει η Κομισιόν κάποιες διευκρινήσεις από αυτό. Μετά όσον αφορά τις εσωτερικές υδάτινες οδούς, ε, βλέπουμε ότι όλη η πρόταση ε, βλέπουμε ότι θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και θα υποβάλω και μια τροπολογία. Κύριε Πρόεδρε, μετά στη συνέχεια είπατε ότι έχετε μόνο μια σελίδα για την γνωμοδότησή σας. Σίγουρα θα υπάρξουν και τροπολογίες που θα υποβληθούν. Στην παραγραφό 9, για παράδειγμα, αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε λίγο χρόνο, χώρο μάλλον, δεδομένου του μιλάει για τουρισμό, μπορούμε να το βγάλουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή στην προηγούμενη ζωή μου ασχολιόμουν με μικροϋπολογισμούς, θέλω να σας πω κάποια πράγματα. Δεν θέλω να αποθαρρύνω τους φίλους μου, αλλά πραγματικά είναι προς συμφέρον μας να είναι εξαιρετικά σαφής η θέση μας. Αν όλοι αρχίσουν τώρα να καταθέτουν τροπολογίες για να για τη διατύπωση, για τα προγράμματα. Θα έχουμε τον κατάλογο για τον Άι Βασίλη, αλλά δεν θα καταλάβει κανεί τίποτα. Θα εξαφανιστεί μέσα στι τροπολογίε το βασικό μήνυμα. Και το βασικό μήνυμα είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που συνδέονται με τον προϋπολογισμό αυτό. Το βασικό δημοσιονομικό μήνυμα ποιο είναι λοιπόν. Πρώτον, οι μεταφορές πρέπει να λαμβάνονται στο σύνολό τους υπόψη στην κατάρτιση προϋπολογισμού γιατί σας είπα, αλλιώ θα χαθούμε μέσα στις τροπολογίες. Καλά κάνατε. Και επανήλθατε στο χρηματοδοτικό μέσο Connecting Europe. Σωστά αυτά που είπατε, αλλά οι χώρες ε, του Ταμείου Συνοχής ε, που επιθυμούν να λάβουν αυτά τα δισεκατομμύρια δεν επιθυμούν να έχουν την κεντρική διαχείριση με την προστέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα. Θέλουν την ελευθερία τους. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο κάποια κράτη στο όνομα της συνοχής έστω θα ήθελαν να μετάσχουν σε αυτό το κίνημα υπέρ της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Το ίδιο δε ισχύει και για τα κράτη που προκρίνει την ανταγωνιστικότητα. Δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε ε, να, την, ε, να κάνουμε αυτό το στρίβιν δια του αραβόνους. Εγώ παίρνω τα δέκα μου και φεύγω και δεν με νοιάζει για την ανταγωνιστικότητα. Πιστεύω ότι Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και κυρίως σοβαρό πρόβλημα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για την ανακατανομή κονδύλιων. Μα η συνοχή τι είναι, δημοσιονομική αλληλεγγύη. Ε, και ε, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ισούται με την κεντρική διαχείριση των κονδυλίων για κάποιους. Όλοι γνωρίζουν ότι το πρόβλημα είναι το όγκος ε, του προϋπολογισμού, δηλαδή τα κονδύλια που θα μας χορηγηθούν μετά τον αγώνα ανάμεσα στα κράτη που δεν θέλουν να πληρώσουν, τα άλλα που θα πληρώσουν, οι άλλοι που ζητάνε σε κάποιους άλλους να πληρώσουν. Και είμαστε σε αυτό το σημείο καμπής, διότι θα συζητήσεις με το Συμβούλιο ήμασταν ε, ε, στον αστερισμό της λιτότητας, ε, αλλά δεν πιστεύω ότι ακόμη και με τις νέες εξελίξεις θα έχουμε μεγάλες παρεκκλήσεις σε σχέση με τα αρχικά προ... τις προτάσεις. Πάντως, Ξαναλέω, όλοι θέλουν να προωθήσουν το πρόγραμμά τους, να πούνε τι τους ενδιαφέρει, τι προτιμούν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, διότι δεν είναι εντελώ ακατάληπτη η πρότασή μας. Ένα άλλο που επίσης με ανησύγησε είναι όταν έμαθα ότι ε, το χρηματοδοτικό μέσο Connecting Europe πήγε στην κατηγορία ΑΑ ανταγωνιστικότητα, ενώ πριν ήταν στο ΑΒ. Μάλιστα. Καλό και αυτό, γιατί θεματικός πώς ταιριάζει καλύτερα, αλλά... Ε, συγγνώμη, αλλά περικόπτουμε και συμπιέζουμε τον προπολογισμό και δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό. Στο κοινοβούλιο δε. Ζητήθηκε και επετεύθη κάποια ζητήματα όπως το GMES να επανέλθουν μέσα στον προϋπολογισμό. Ε, συμφώνησαν όλοι, συμφώνησαν για το ίδιο δημοσιονομικό κονδύλι. έξω και το πρόβλημα, γιατί θα ε, συνιστά αυτό μεγάλη απειλή για μας, για τους λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ιάλισεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το όσα είπε ο κύριος ε, Μακένη, ήθελα καταρχώς να συγχαρώ εσάς ε, διότι συγκεντρώνοντας όλα αυτά τα μέσα καταφέρατε να εντοπίσετε όλα τα προβλήματα παρότι στην παρουσίασή σας προσθέσετε και κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες. Ε, δεν ε, παρέχονται όμως κάποια ελάχιστα ποσά για τη χρηματοδότηση αυτής της νέας δέσμευσης για τα κονδύλια υποδομών με πραγματική προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Διαφορετικά δεν υπάρχει, δεν έχει νόημα όπως ε, εάν έχουμε τέτοιε περικοπές Θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες μας πού θα κάνουμε τις περικοπές, τι θα μειωθεί ή το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεργαστεί βάσει τις θέσεις που υιοθέτησε μέσα στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα και να πει ότι αν πέσω κάτω από αυτό που θεωρούμε ζωτικό ελάχιστο, τότε το Κοινοβούλιο απλά θα απορρίψει ε, αυτό που θα καταλήξει να είναι μια αστεία πρόταση. Δηλαδή πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι το οποίο θα μας κάνει τον περίγελο της δημόσιας γνώμης, της κοινή γνώμης. Έχουμε εδώ την Κομισιόν και θα πρέπει να πιστεύω να τους ρωτήσουμε πως αυτοί αντιλαμβάνονται αυτή την κίνηση που υπάρχει στην επικεφαλίδα 1α ε, φυσικά υπάρχουν κάποια έργα όπως το Γαλλίο που μας ενδιαφέρουν, αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί. Όχι μόνο κίνδυνος των λιγότερων κονδυλίων, ε, Πιστεύω ότι όσοι υπερασπίζονται αυτή την επικεφαλίδα έχουν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι αν έχουμε αυτά τα 10 δι από το Ταμείο Συνοχής ε, για το σύνολο τη δουλειά μα. θα βρεθούμε ενώπιον μια κατάσταση όπου ο καταμερισμό θα γίνει με τρόπο που δεν θα είναι, θα είναι Θα θέλαμε λοιπόν να μα πει η Κομισιόν ποια είναι η στρατηγική τη ε, προ υπεράσπιση αυτή τη προσέγγιση. Αναφέρθηκε ότι στο ERTF ε, υπάρχουν σημεία τα οποία θα μπορούσαν να μελετηθούν και υπό όρους μεταφορών. Εδώ δεν μιλάμε απλά για αποκέντρωση της ε, διαχείρισης. Όσον αφορά την ε, προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και το μορφή που το Ταμείο το στο μέλλον, Χρειαζόμαστε ποιοτική υλοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόσο για τον τουρισμό επίσης έχετε δίκιο εφόσον έχουμε την νομική βάση. Για πολύ καιρό έλεγε ο κόσμος ότι δεν υπήρχε προπολογισμό, δεν υπήρχε ικανοποιητική νομική βάση και ξαφνικά ο προπολογισμό έχει εξαφανιστεί λέει το Κοινοβούλιο. Αυτό τη μάχη θα πρέπει να το δώσουμε. Διότι αυτά τα προγράμματα μπορεί να μας βοηθήσουν να ξανεντάξουμε κάποια σχέδια, είναι προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, ο κ. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως η κυρία Ελεζάνδρ και διαφορετικοί μελητές έχω μια ερώτηση προς την Κομισιόν αλλά και γενικότερη φύση ερώτηση όσον αφορά τα ζητήματα που αναφέρει η κυρία Μάισνερ και ο συνοδελφός μου Πίτερ Βαντάλεν αφορά τα όσα ε, ανέφερε ως μόχλευση κύριε ε, Μάισνερ. Το έχω μελετήσει το ζήτημα ειδικότερα όσον αφορά το μηχανισμό Connecting Europe. Στο πλαίσιο αυτού λοιπόν η όλη ιδέα των ε, ομολόγων προγραμμάτων για πιλωτικά προγράμματα και μου λένε οι συναδελφοί μου στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ότι στόχος αυτών των ομολόγων θα είναι να αποκομιστούν 80% από τον ιδιωτικό τομέα με το 20% να χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Ε, θα, θα, ήθελα λοιπόν να μας πει καταρχάς η Κομισιόν την απόψή τη για αυτό το ζήτημα και το δεύτερο που θα ήθελα να μάθω είναι τι θα συμβεί κύριε Πρόεδρε εσείς θα θυμάστε εσείς εγώ και ο Μάρτιν Κρόσιος να είμαστε οι μόνοι που θα θυμόμαστε ότι όταν αρχικά είχαμε ξεκινήσει το πρόγραμμα TEN για να συμπεριλάβουμε το πρόγραμμα Καλλιλέο τότε η Κομισιόν είχε πει δεν θα δοθούν χρήματα ε, από το τένις για τον Γαλιλαίο πάνω από 20% και μετά μας είπαν ο ιδιωτικός τομέας δεν θέλει να εμπλακεί συνεπώς χρειαζόμαστε περισσότερο ποσοστό για να χρηματοδοτήσουμε τον Γαλιλαίο. Αυτό που θα ήθελα να μου πείτε, τι διασφαλίσει έχουμε αυτή τη φορά από την Κομισιόν, ότι οποιαδήποτε προγράμματα που υποτίθεται ότι θα προσελκύσουν 80% ιδιωτικέ επενδύσει, είναι διασφαλισμένο ότι θα τα πραγματοποιήσουν αυτά και ότι δεν θα ξαναέρθουν σε εμά να μα ζητήσουν χρήματα από ήδη υπάρχοντα προγράμματα για να τα χρηματοδοτήσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση θα μπει στο παράρτημα της ενδιάμεσης έκθεσης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που θα αναμένεται να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Αναμένεται επίσης μια απόφαση σχετικά με τα κονδύλια που θα διατεθούν για τον επόμενο πλαίσιο 2014 ως 20. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που θα παγιοποιήσουν τη θέση του Κοινοβουλίου ε, και ως εκ τούτου και την εντολή της διαπραγματευτικής ομάδας ε, προτού λάβει χώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα συμφωνήσω πως ε, η έκθεση δεν πρέπει να τροποποιηθεί ως προς την ουσία της, πλην όμως θα πρέπει να προσθέσουμε κάποια στοιχεία. Πρώτον, Οι δράσεις για τον τουρισμό και για τις μεταφορές ε, θα πρέπει να, συμπερι... να παραμείνουν στα κεφάλαια όπου βρίσκονται τώρα. Μήπως θα έπρεπε να προσθέσουμε κάποιες ε, γενικόλογες αναφορές ε, σε σχέση με το χρηματοδοτικό μέσο Connecting Europe. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση πάντως ότι θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες για οποιοδήποτε πρόγραμμα. Στην έκθεσή μας υπάρχουν στοιχεία που υπάγονται στη διαδικασία, συνήθως νομοθετικής διαδικασίας. Ε, γι' αυτό Προτείνω να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση, διότι έτσι θα εξασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό επίπεδο χρηματοδότησης για τα προγράμματα που σχετίζονται με τις μεταφορές. Είτε βασιστούμε στην πρόταση της Επιτροπής, είτε στην έκθεση της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Μόνο έτσι θα είναι πλήρη η έκθεσή μα και θα έχουμε μια ε, ξεκάθαρη εικόνα για το επόμενο πλαίσιο, 2014 ως 20. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη διότι έχασα την αρχή της συζήτησης μόλις έφτασα. Φαντάζομαι ότι θα έχουν γύρει τα ίδια ζητήματα πολλοί συνάδελφοι. Θα επαναλάβω μόνο τα εξή. Οφείλουμε να έχουμε επίγνωση του κινδύνου που διατρέχουμε και στην προκειμένη περίπτωση οι επενδύσεις για την περίοδο 2014 2020 τα ε, η έρευνα, τα αναπτυξιακά ταμεία θα πέσουν θύματα στο βωμό της, ε, του συμβιβασμού ανάμεσα ε, στους καθαρούς εισφορείς και στους καθαρούς δικαιούχους που είναι φυσικά οι οι χώρες του Ταμείου Συνοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο αποστείλει ένα σαφές μήνυμα ότι δηλαδή για να διασφαλίσουμε μια εύρωστη οικονομία για τα επόμενα έτη χρειαζόμαστε αυτή την χρηματοδότηση και θα πρέπει τα προγράμματα μεταφορών να αναδειχθούν σε προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι ε, αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το συζητήσουμε με συναδέλφου και από άλλε επιτροπέ. Επίση, θα ήταν χρήσιμο να μα δώσει πολεμοφόδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μα πει Πιο συγκεκριμένα, ε, ποιες είναι αυτές οι επενδύσεις που θα μας εξασφαλίσουν μια πιο ταχύ ρυθμή ανάπτυξη. Ποιες επενδύσεις θα πρέπει να προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να αποφασίσουμε πώς πρέπει να κινηθούμε για το μέλλον. Ενδεχομένως θα μπορούσατε να μας δώσετε στοιχεία για τις προηγούμενες επενδύσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πακέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως ε, πιστεύω ότι το σχέδιο έκθεσης ε, καλύπτει όλα τα ε, βασικά στοιχεία των προκλήσεων που αντιμετωπίσουμε στον τομέα της χρηματοδότησης των μεταφορών σε συνδυασμό το με το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Ε, η φιλόδοξη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την, ε, το χρηματοδοτικό μέσο Connecting Europe βασίζεται στα μέχρι τούδε αποτελέσματα αλλά και στα αυτά αποτελέσματα που αναμένουμε από αυτά τα προγράμματα και γι' αυτό ισχυριζόμαστε ότι όντω αυτή η χρηματοδότηση είναι ελάχιστη δυνατή και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σα ω προς την αρχική μας πρόταση, ω προ τα 10 δις του Ταμείου συνοχή που θα εισαχθούν ε, στο ΣΕΦ. Ε, πολλοί ε, προλαλήσαντες σχολίασαν αυτό το ζήτημα και σωστά είπαν ότι ο στόχος είναι να αποκομίσουμε τη τη δυνατή ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία από τη χρηματοδότηση και τίποτε άλλο και πιστεύουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί συμπληρωματικά προφανέστατα με την αυξημένη χρηματοδότηση βάσει διαφόρων μέσων της περιφερειακής πολιτικής μεταξύ των οποίων και το Ταμείο Συνοχή. Ε, στην εισαγωγή που κάνετε για την έκθεση αναφερθήκατε και στο πρόγραμμα Μάρκο Πόλο και σωστά αναφέρατε ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει τώρα να το Πάρκο Πόλο να μπει στι υπηρεσίε μεταφορά εμπορευμάτων. Λοιπόν, η επιλογή μα βασίζεται σε δύο στοιχεία. Πρώτον, streamlining και απλούστευση για όλα τα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά εξίσου σημαντικό είναι το εξή ε, να προσφέρουμε νομική βάση και πλαίσιο για την κατάρτιση πολιτική ω προ την ανάπτυξη υποδομών, ούτω ώστε να καλυφθούν και οι υπηρεσίε που θα προσφέρονται χάρη σε αυτήν την ε, νέα υποδομή και Πέρα από το βασικό δίκτυο, λοιπόν, θα πρέπει να προγραμματίσουμε, να σχεδιάσουμε μαζί την υποδομή σε μια πρώτη φάση και τις υπηρεσίες στη συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο ε, θέλουμε τα μέτρα τύπου Μάρκο Πόλο να συνδεθούν με το χρηματοδοτικό μέσο ΣΕΦ. Τέλος... Ε, είναι η ελάχιστη δυνατή χρηματοδότηση όντω, <coughs> αλλά θα πρέπει να τη συνδυάζουμε και με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά ούτω ώστε ε, να γίνουν με λογικό τρόπο τα επόμενα έτη ε, οι μεγαλύτερες δυνατές επενδύσεις για τα TEN-T. Ε, ο κύριος Βαντάλεν ρώτησε για το Σενέσκο. Το πρόγραμμα ε, στη Γαλλία έχει απασχολήσει πολύ τον τύπο αυτό το θέμα. Το Γαλλικό Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος ε, και πέρα από τα δημοσιεύματα ε, και βάσει της έκθεσης ε, του Αρμοδίου Υπουργείου δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Πάντως αυτό το πρόγραμμα θα συμπεριληφθεί στο γενικότερο σχεδιασμό των υποδομών στην Ευρώπη. Η κυρία Σαγέλα Σέντερ η ερώτηση σχετίζεται με τις κατηγορίες. Είναι στο 1α ή στο 1β. Κοιτάξτε, προτείναμε αλλαγή κατηγορία προτείναμε ε, το 1β όντω, Ταυτόχρονα όμως ε, η πρόκληση του να διατηρηθεί δηλαδή το ΣΕΦ ε, είναι μεγάλη όποια κατηγορία και αν επιλέξουμε τα κράτη που θεωρούν ότι δεν είναι επαρκή σε η και τα, οι βουλευτές του Κοινοβουλίου που πιστεύουν το ίδιο πράγμα θα πρέπει να ε, προτάξουν ευλόγα επιχειρήματα τόσο ώστε να καταδείξουν πως οι επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών ε, θα καρποφορήσουν περισσότερο να συνδυαστούν με ε, την ΣΕΦ, το χρηματοδοτικό μέσο ΣΕΦ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πακέλε, κύριο Σίμψον. Θα ήθελα τώρα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Ξέρω ε, μάλλον, όπως σας είπα, είμαστε περιορισμένοι ως προς το μέγεθος ε, της έκθεσης ε, σε μία σελίδα και αντί να περάσουμε αμέσως στη συζήτηση με τους σκιώδεις και να καταλήξουμε σε πολλές τροπολογίες. Θέλω να προσέξουμε αυτά που είπαν συνάδελφοι όπως ο Ντομινίκ Ρίκε. Δεν μπορούμε να επιδιώκουμε τόσες πολλές τροπολογίες ώστε να αποδυναμώσουμε τελικά το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Μην ξεχνάτε συνάδελφοι επίσης ε, ότι ε, αυτό συνδυάζεται με τη συνολικότερη ε, δράση του Κοινοβουλίου στην διαπραγματευτική ομάδα και σε όλες τις συναρμόδιες επιτροπές. Ποια είναι η στρατηγική λοιπόν που γενικώ ακολουθείτε, όπου μπορούμε δεν αποκλίνουμε ε, σε μεγάλο βαθμό από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αναμένεται μάχη με το Συμβούλιο για κάποιο ζήτημα. Λοιπόν, αυτή η μάχη πώς θα ε, εξελιχθεί, ε, θα εξελιχθεί αφού το Συμβούλιο δηλώσει πού θέλει να γίνουν οι περικοπές. Ε, μετά θα αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε. 10 Ιουλίου είναι η ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών. 18 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών και μετά το καλοκαίρι έχουμε χρόνο ακόμη για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε ποια θα είναι η γραμμή δράσης μας. Στις 18 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί η έκθεση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών Θελημένη όρισε αυτήν την ημερομηνία, ούτω ώστε να συντονιστούμε με τη λήψη αποφάσεων του Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, μόλι ε, ε, μάθουμε τη θέση του Συμβουλίου, θα περάσει το θέμα στην Ολομέλεια το Νοέμβριο, όταν θα έχουμε δηλαδή την τελεσίδικη θέση του Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστούμε και πάμε στο επόμενο σημείο. Ταμείο τα Ταμείο ανάπτυξη τη Υπέθρου. Έχουμε τρεις διαφορετικές εκθέσεις, Μάικλ Κράμερ. Καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδει εισηγητές. Είχαμε καλή συνεργασία και σε κάποια σημεία καταφέραμε να βρούμε και συμβιβασμούς. Ε, το συνολικό πακέτο αποτελείται από τρεις ε, γνωμοδοτήσεις. Ε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες για όλα τα ταμεία, κανόνες για το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης. Εμένα με ενδιαφέρει η πτυχή των μεταφορών και στις τρεις αυτές γνωμοδοτήσεις. Υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν γενικά με τα ταμεία, αλλά έχω εξετάσει ε, την πτυχή των μεταφορών. Διότι οι άλλες πτυχές εξεταστούν από τις άλλες επιτροπές. Έχουμε λοιπόν τον γενικό κανονισμό και καταφέραμε ε, στο 9-1-7 να καταλήξουμε σε συμβιβασμό με κοινή διατύπωση και για τις ε, τρεις πτυχές. Αποτελεσματικότητα, commodality και αποτελεσματικότητα περιβαλλοντική. Βλέπω ότι αυτοί που συμμετείχαν χαμογελάνε και χαίρονται με το συμβιβασμό που βρήκαμε. Μιλάμε για περιφερειακές, τοπικές και αστικές μεταφορές και λείπουν οι υπαίθριες. Κάποιοι πιστεύουν ότι στις περιφερειακές και αστικές ε, συμπεριλαμβάνονται και οι υπαίθριες. Αλλά θα ψηφίσουμε πάνω στο θέμα αυτό. Στο σημείο αυτό δεν καταφέραμε να βρούμε συμβασμό στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, βρήκαμε και εδώ κοινή διατύπωση. Ιδιαίτερα ε, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή των νέων κρατών μελών. Θέλουμε μείωση της ε, ηχορύπανσης ε, και έχουμε πει στην Κομισιόν ότι είναι δυνατόν να τεθούν συγκεκριμένε προϋποθέσεις. Ε, θέλουμε να τις καθορίσουμε και ξέρουμε ότι το παράρτημα με τους δείκτες απειλείται να διαγραφεί. Δεν έχουμε συμφωνήσει σχετικά με το τι είδους ε, επενδύσεις για τις μεταφορές είναι δυνατές. Ε, θα πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε μόνο αηφόρες επενδύσεις. Ε, ο κύριος Σερικέ θεωρεί ότι όλες οι επενδύσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Δεν καταφέραμε εδώ να καταλήξουμε σε συμβασμό. Θα πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε. Όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής, μας ενδιαφέρει εδώ η συνέπεια με τον γενικό κανονισμό. Μας ε, ενδιαφέρουν ε, τα διάφορα είδη μεταφορών, ε, μείωση των, της χορύπανσης και περαιτέρω ανάπτυξη των σχετικών δικτών. Ε, σημαντικό πρόβλημα είναι τα διασνοριακά σημεία. Πριν ε, πολλά χρόνια θέλαμε να έχουμε ένα γενικό δίκτυο. Τελικά έχουμε καταλήξει σε μια λύση patchwork και ε, υπάρχουν στα σύνορα πάντα σημεία προβληματικά. Προσλέπω στην καλή συζήτηση και στην ψηφοφορία αύριο. Ε, και ευχαριστώ όλους ε, τους ε, σκιώδεις συζητητές για την επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ Μάικλ, ο κύριος Ρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ στη μία έκθεση όπου είμαι σκιώδης εισηγητής. Οι συνάδελφοί μου θα αναφερθούν στις άλλες. Σημαντικό για μένα είναι ότι ο εισηγητής κατά τη γνώμη μου έχει φτιάξει μια καλή έκθεση, έχει πολύ καλές προϋποθέσεις, έχει συμπεριλάβει πολύ καλές προϋποθέσεις και Αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στην ε, έκθεση αυτή θα πρέπει να περιοριστούμε ε, στο θέμα των μεταφορών ε, και όχι να απορρίψουμε το σύνολο της περιφερειακής πολιτικής. Θα μπορούσαμε άλλωστε μέσω της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης να ρυθμίσουμε κάποια επιμέρους θέματα αν είναι απαραίτητο. Θέλουμε εδώ να τονίσουμε κάποια θέματα που αφορούν τις μεταφορές Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η έκθεση του κυρίου Κράμερ είναι κάπως πιο πράσινη. Εμείς ε, προσπαθήσαμε με ε, τροπολογίες ε, να συμπεριλάβουμε και άλλες πτυχές, αλλά σημαντικό για μένα και στη συζήτηση ήταν ότι πριν ένα χρόνο θέσαμε τον γενικό προσανατολισμό. Ο Επίτροπος Χάνη είπε τότε ότι αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε προϋποθέσεις ε, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. θα πρέπει λοιπόν να εξεταστούν ε, οι πτυχές που αφορούν ιδιαίτερα τις μεταφορές ε, σε διάφορα σημεία. Έχω υποδείξει και μάλιστα ο εισηγητής ε, έχει αλλάξει τα σχετικά σημεία. Ε, σημαντικό είναι να μην μπλοκάρετε ένα καλό έργο γι' αυτό. Ε, δεν θα πρέπει να χάνουμε και την ε, σχέση με άλλα προγράμματα όπως το Natura 2000. Όσον αφορά την τροπολογία 91, ε, συμφωνώ απόλυτα με το περιεχόμενο, δεν ξέρω όμως εάν η πτυχή που αναφέρεις εδώ έχει τη θέση της εδώ. Αν κάθε επιτροπή ε, θέλει να συμπεριλάβει τις δικές της λεπτομέρειες, αυτό ίσως είναι υπερβολικό. Ε, εδώ δηλαδή διαφωνεί το ΕΛΚ όχι όσον αφορά το περιεχόμενο αλλά με τη θέση της τροπολογίας αυτής. Τέλος ε, θα ήθελα να πω ότι είχαμε εσωτερικά μια συζήτηση Ε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις τροπολογίες 46 και 132. Υπάρχει η διευκόλυνση Connecting Europe Ε, πιστεύω ότι θα, όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης ε, θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο για να έχουμε συζητήσεις ε, με τις αρμόδιες επιτροπές. Αυτό όμως ε, δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε και να δώσουμε σαφεί απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα των ε, χωρών ε, συνοχής. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και ελπίζουμε αύριο να έχουμε καλό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον κύριο Κράμερ να εκπονεί έκθεση που να μην είναι πράσινη. Η κυρία Σελαλόβα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήμουν σκιώδης για τις τρεις αυτές εκθέσεις και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να τις σχολιάσω από κοινού. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Κράμερ ε, για την ε, ιδιαίτερα ένεργο συμμετοχή του και τις τροπολογίες του θεωρώ ότι είναι επιτυχημένες οι προσπάθειες που κάναμε. Η συμβαστική λύση της Επιτροπής Ρέτζη δείχνει με σαφήνεια ποιες είναι οι προτεραιότητες κατά τη γνώμη της Επιτροπής Μεταφορών, ποιες πρέπει να είναι οι βασικές επενδύσεις στο μέλλον κατά τη γνώμη μας για τα διαρθρωτικά ταμεία, για το περιφερειακό ταμείο, ταμείο αγροτικής ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Χρειαζόμαστε φιλική ως προς το περιβάλλον υποδομή για την καταπολέμηση της συμφόρησης σε όλα τα είδη μεταφορών, είτε είναι πλωτές, είτε οδικές, είτε είναι αέριες, ε, γιατί τον εξυγχρονισμό της υποδομής ε, θα πρέπει να εξετάσουμε την προσέγγιση πολυτροπικότητας. Έχουμε την πράσινη βίβλο για τις μεταφορές, στο οποίο μπορούμε να βασίσουμε ε, την θέση μας σε όλα τα έγγραφα που έχουν εκπονηθεί σχετικά με τα προγράμματα TNT καθώς ε, και το κομμάτι της συνοχής ε, στην ε, στρατηγική 2020 για πιο συγκεκριμένα την αρχή του ότι ο Ριπένων πληρώνει. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καθαρές μεταφορές και στην Ήπεθρο και στις αστικές περιαστικές περιοχές. Θεωρούμε πως οι βασικοί αποδέκτες ε, των επιδοτήσεων ε, πρέπει να είναι αυτοί που βρίσκονται ε, στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές η επανάπτυξη αυτών των περιοχών έχει ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό αποδίδουμε έμφαση σε αυτό το σέμα. Θέλουμε λοιπόν τα εναλλακτικά σενάρια που θα επιλέξουμε να εξυπηρετούν τους πολίτες ε, για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ε, στις μεταφορές μας. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω την υποστήριξή σας επ' αυτού για μια προφορική τροπολογία σχετικά με την αρχική τροπολογία 125 Επίσης, συμπληρωματική τροπολογία αντί για το ε, ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ως προς τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Ε, ένα λιγότερο αμφιλεγόμενο θέμα ήταν η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να εμποδίσει τις δημόσιες επενδύσεις σε κάποιες περιοχές. Δεν είμαστε υπέρ αυτής της πρότασης στην ομάδα μου, διότι Ε, αυτός ο τρόπος ε, μεταφορών ε, είναι εξίσου σημαντικός είτε μιλάμε για πολύ αναπτυγμένες περιοχές είτε για λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Σας περάσω τώρα στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Είναι κέρια σημασία η συζήτηση σχετικά με την λειτουργία αυτού του μέσου. Γι' αυτό το λόγο θα υποστηρίξω τις τροπολογίες που θα μας οδηγήσουν σε εντατικότερο διάλογο για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την Επιτροπή για την Επικοδομητική Συνεργασία τους και είμαι ε, σίγουρη ότι θα βρούμε και ε, λύσεις για τις σημαντικές τροπολογίες. Ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη για το κρύωμα που με ταλανίζει ίσως αυτός ο αντιευρωπαϊκός άνεμος που φυσάει από όλες τις πλευρές φταίει. Θα είμαι λοιπόν σύντομος. Επιτεύχθηκαν διάφοροι συμβιβασμοί στους οποίους δεν χρειάζεται να σταθώ περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτούς. Είναι ειρηνικοί. Παρότι αρκετά συγκεντρωτική, αρκετά πράσινη μάλιστα. Αλλά φυσικά θα δώσει την πινελιά του ο εισηγητής στο κείμενο αυτό. Και τι συμμερίζομαι. Όσον αφορά κάποιες άλλες τροπολογίες, ωστόσο, η ομάδα Άλντε δεν συμφωνεί κυρίως ε, εξαιτίας του γεγονότος ότι πρόκειται για τροπολογίες ε, φύσης τέτοιας που ε, που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν καλύτερα από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως η εκ των προτέρων αρεσιμότητα, η εκ των υστέρων αρεσιμότητα, η μακροοικονομική αρεσιμότητα, οι περιφέρειες ζητήματα που συζητήθηκαν ήδη γνωρίζουν καλά οι συναδελφοί από την Επιτροπή Ανάπτυξη για το τι μιλάω. Ήθελα να αναφερθώ αντιθέτω σε κάποιε τροπολογίε ώστε να πω ότι υπάρχουν κάποιες, κάποια ερωτήματα για τα, στα οποία η Επιτροπή Μεταφορών όπως έλεγε και ο συνάδελφος Γκρόστα θα πρέπει να σκεφτεί περισσότερο το ένα αφορά τον κανονισμό για τι κοινέ διατάξεις, ειδικότερα το μηχανισμό συνδέεται στην Ευρώπη το Connecting Europe και ειδικότερα το γεγονός ότι 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής ε, θα μετατοπιστούν και κάποιες τροπολογίες ε, όπως η 135 όπου ζητείται το ποσό χρηματοδότησης ε, να δοθεί σε ίδια ποσόστοση από την Κομισιόν. Εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτό και θα ψηφίσουμε κατά αυτής τροπολογίας 135. Επίσης είμαστε αντίθετοι με την τροπολογία εκείνη που προβλέπε μεταφορά του ποσού που αφορά τα κράτη-μέλη που έχουν δικαίωμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής που συναποφασίζεται. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιλέξει η Κομισιόν όσον αφορά τα προγράμματα που έχουν παρουσιαστεί ερμηνεύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συνολικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το συμφέρον επιμέρους κρατών μελών που όπως γνωρίζουμε ε, προσπαθούν να απαιτήσουν πολλές φορές ε, φυσικά δικαίως ε, ζητήματα ειδικού χαρακτήρα. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα και κάποια άλλα ερωτήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ολοκληρώσω εδώ διότι αφορούν απλά μεμονωμένες τροπολογίες. Τέλος, ήθελα να πω ότι το Άλντε θα ψηφίσει κατά της τροπολογίας που αφορά φορά τον κανονισμό ο οποίος προβλέπει στην ενδιαμισία θεώρηση των κονδυλίων που εκορούνται σε προγράμματα που έχουν επιλεχθεί με την αρχή ο πρώτος που φτάνει εξυπηρετείται πρώτος εκεί θα ε, ψηφίσουμε αρνητικά. Ευχαριστώ. Roberts. Κύριε Ζήλα Ρόμπερτ. Θα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάικλ για το ε, προσπάθειά του να επιτύχει συμβιβασμού στο σύνολο υπάρχουν βρίσκουμε περισσότερα θετικά σημεία παρά Όσο τα, όσον αφορά τα κονδύλια, θα υποστηρίξουμε τις συμβαστικές G και I για τα δίκτυα μεταφορών. Και μετά τη CEF ε, για το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη. Για το γενικότερο κανονισμό, για τις διατάξεις εδώ, Ένα πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αυτό το νέο όριο, το κατόφλι για κάποια νέα κράτη-μέλη, το 2,5 δηλαδή του ΑΕΠ, οδηγεί σε πολιτική αβεβαιότητα. Και τα κράτη-μέλη θα ήθελαν να έχουν και τα 10 δισεκατομμύρια στο εθνικό αυτό ποσό. Ο Επίτροπος Κάλλας το φθινόπορο, παρουσίασε τη διευκόλυνση Connecting Europe, ενώνοντας την Ευρώπη. Ε, εξήγησε λοιπόν ότι αυτά τα 10 δισεκατομμύρια ε, θα πρέπει να θεωρηθούν προσθήκη, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου. Και επίση, όταν ένα κράτο κράτος μέλος ε, φτάσει το κατόφλι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνει πια καμία χρηματοδότηση. Επίσης, ε, θα ήθελα να πω ότι τα 10 δις ε, της διευκόλυνσης Connecting Europe είναι μια προσέγγιση ε, της Κομισιόν είναι ένα είδος benchmarking ε, ε, για τα κράτη-μέλη. Όταν ένα κράτος μέλος δεν εξαντλήσει τους πόρους, τότε μπορούν άλλα κράτη-μέλη να επωφεληθούν από τους πόρους αυτούς. θα χαιρόμουν εάν η Επιτροπή στηρίξει τουλάχιστον μέρος της πρότασης αυτής. Ευχαριστώ κύριο Ζρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα παρέμβω μόνο για το κομμάτι για το, με το οποίο ασχολήθηκα εγώ, δηλαδή με το Ταμείο Συνοχή. Ήθελα να ευχαριστήσω κατάρχο τον Μάικλ για την ευχάριστη συνεργασία που είχαμε, την ευκολία στην επαφή και στη συζήτηση. Συμφωνήσαμε πιστεύω σε πολλά σημεία συμπεριλαμβανομένου συμπεριλαμβανομένης και μιας διαφωνίας που αντιστοιχεί σε ανησυχίες πραγματικές που έχουμε όλοι. Δεν συμφωνήσαμε αντιθέτως για την αιρεσιμότητα όσον αφορά τα, προγράμματα, τα δικά προγράμματα στο πλαίσιο του Ταμείου συνοχή. Αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα διότι σε αυτήν την Επιτροπή προτιμάμε να υπερασπιζόμαστε έργα προστιθέμενης περιβαλλοντικής αξίας και γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη συχνά έχουν την τάση να πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση ε, δεδομένου ότι δεσμεύουμε 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής για το πρόγραμμα συνδέοντας στην Ευρώπη εάν προσθέσουμε μια αιρεσιμότητα επιπλέον όσον αφορά τα οδικά έργα στο πλαίσιο του Τέμιου ε, Αυτό παραπάει και μετά έχουμε δύσκολες συζητήσεις περίπλοκες με κάποια κρατημέλη επί του θέματος. Ε, δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για τα θέματα της αιρεσιμότητας όσον αφορά τα δικά έργα. Στα υπόλοιπα συμφωνήσαμε. Ωραία, ο κύριος Μαϊνέσκου. Ευχαριστώ για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπου είμαι σκιώδης εισηγητής. Θα ήθελα να πω μόνο πως συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με τον κύριο Κράμερ και έχει μια πράσινη οικολογική πτυχή στο χαρακτήρα του, από ό,τι μας λέει. Δυσκολευτήκαμε να καταλήξουμε σε συμβασμό, αλλά ε, τα καταφέραμε τελικά. Σχετικά με τον τουρισμό, συμφώνησε ο κύριος Κράμερ ότι πρέπει να έχουμε ξεχωριστό κεφάλαιο για τις μεταφορές. Πολύ θετικό αυτό. Αν κρίνω τώρα από την τωρινή μορφή της έκθεσης ε, και φυσικά θα κρίνουμε και από την έκβαση της ψηφοφορίας, ε, ε, θα έλεγα ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Επιτροπή των Μεταφορών και η τελική έκθεση θα έπρεπε να συμπεριλάβει διάφορες από αυτές τις παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε η κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Κράμερ ε, για τις προσπάθειες που έκανε για να καταλήξει σε συμβαστική λύση. Αληθεύει ότι ε, κατέθεσα διάφορες τροπολογίες ε, και είδα στον κατάλογο ψηφοφορίας ότι οι συγκεκριμένες τροπολογίες δεν υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Μεταφορών. Μιλώ συγκεκριμένα για τον κατάλογο των πόλεων που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να προσδιορίζει τον των προτέρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σχετίζονται και με τις ημερομηνίε, τις προθεσμίες που προβλέπονται για την έγκριση διαφόρων εγγράφων από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα τώρα να συναντηθώ και πάλι με τους συναδελφούς σκιώδης εισηγητές ε, για να δούμε αν θα ε, μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβασμό με την Επιτροπή Ανάπτυξης, ε, διότι πιστεύω πραγματικά ότι οι τροπολογίες αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθούν και θα πρέπει να είναι ώστε το δυνατόν πιο σύντομες ε, γίνεται, ούτω ώστε τα, όλα τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν τους ε, κανόνες ε, και τα κριτήρια που θα είναι εφαρμοστέα μελλοντικά, αλλά να το γνωρίζουν, ε, να το μάθουν το ταχύτερο δυνατόν. Ε, γι' αυτό σας μίλησα για τις προθεσμίες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να εκπονήσει τα έγγραφα και να θέσει στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων μερών της πληροφορίε αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ταχύτερο δυνατόν. Για το χρηματοδοτικό μέσο ΣΕΦ προτείνω εθνικά κονδύλια. Θα ήθελα ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό να διοχετευτεί από το Ταμείο Συνοχής ε, για τις υποδομές μεταφορών, όμως χρειαζόμαστε και το σωστό τρόπο, το σωστό μεθηματικό τύπο, διότι οι χώρες ε, που υπάρχονται στα κριτήρια συνοχής ε, δεν θα πρέπει να απολέσουν οποιοδήποτε κομμάτι χρηματοδότηση έχουν στη διάθεσή τους αυτή τη στιγμή και σας σταματώ τώρα, πολύ ωραία. Θα, θα ακούσουμε συγγνώμη, την κυρία Μάιλεν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. Σα ευχαριστώ πολύ από πλευρά τη ε, Κομισιόν. Επικροτούμε τα σχέδια γνωμοδοτήσεων και την αναλυτική δουλειά που έχει γίνει, ιδιαίτερα από τον εισηγητή. Σημειώνουμε τις προτινόμενες τροπολογίες και θα θέλουμε να σχολιάσουμε κάποιες από αυτές. Καταρχήν όσον αφορά τον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις. Στηρίζουμε την υποστήριξη προς ε, μια ε, λυσιτελή προσέγγιση και δεχόμαστε ότι υπάρχουν ε, και κάποιες τεχνικές προσαρμογές όσον αφορά κάποια ποσά. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε περαιτέρω. Όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, πιστεύουμε ότι πολλά από τα στοιχεία αυτά που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη ήδη έχουν ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα στο άρθρο 8 του κανονισμού ε, κοινών διατάξεων ε, και στα άρθρα 87 και 114. Ωστόσο, η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να εξετάσει το θέμα αυτό περαιτέρω. Επίσης, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Φαίνεται να υπάρχει ένα γενικό οριζόντιο θέμα όσον αφορά τις προθεσμίες ε, σε κάποιες επιστροπολογίες, ιδιαίτερα για τις ε, κατεξουδότηση πράξεις, διότι είναι σημαντικό για την Επιτροπή να έχει αρκετό χρόνο για εσωτερικές διαβουλεύσεις και εσωτερικές διαδικασίες. Και γι' αυτό μας ανησυχούν κάπως ε, κάποια πολλά σφιχτά χρονοδιαγράμματα, κάποιες πολύ σφιχτές προθεσμίες που προτείνονται στις τροπολογίες όσον αφορά τον ε, κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, συμπεριλαμβάνονται πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τις ε, προτεραιότητες και πιστεύουμε ότι υπερβολικός βαθμός ανάλυσης ε, στις προτεραιότητες επενδύσεων μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα ερμηνείας και πιστεύουμε ότι αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να είναι γενικοί στόχοι και όχι μακρύς κατάλογοι δράσεων. Σημειώσαμε επίσης την πρόταση οι μεταφορές ε, να μεταφερθούν από τον θεματικό στόχο 7 στον θεματικό στόχο 4 και αυτό μας ανησυχεί διότι πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποσπάσει πόρους από την ε, ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επίσης είναι πολύ σημαντικά. Επίσης έχουμε ε, σημειώσει την συμπερίληψη του τουρισμού και πιστεύουμε ότι καλύτερο θα είναι να μην αναφέρονται συγκεκριμένοι τομείς. Ο τουρισμός είναι συγκεκριμένος τομέας και μπορεί να καλυφθεί από διάφορους ε, θεματικούς στόχους και γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στον κανονισμό. Όσον αφορά τους κοινού ε, δείκτες, ε, επικροτούμε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να τους βελτιώσουμε και είμαστε ανοιχτοί προς συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής. Έχουμε σημειώσει τη συμπερίληψη ε, της κοινωνικής στέγασης σε μια από τις τροπολογίες ε, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ήδη αντιμετωπίζεται, ε, το οποίο ήδη καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Υπέθρου, Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ERDF και πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να γίνει στο, στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Όσον αφορά τον τουρισμό και το Ταμείο Συνοχής, θα θέλαμε να τονίσουμε το γεγονός ότι η, η συνθήκη δεν δίνει ρόλο ε, στον τουρισμό στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μας ε, για κάποιες από τις τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάικλ. Έχεις κάτι να προσθέσεις? Ναι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για ε, τη συζήτηση και για τους επένους για τη δουλειά μου. Δεν το έχουμε συνηθίσει ε, Ω πράσινοι, αλλά με λίγη προσπάθεια καταφέρνουμε να βρούμε συμβιβασμού που να καλύπτει και τους ε, ε, και, και τις άλλες πολιτικές ομάδες. χαιρόμαστε λοιπόν και εσύ μπορείς να χαίρεσαι. όσον αφορά τα 10 δις και αυτό που είπε ο Ματιό Γκρός και θα, θα πρέπει να συζητήσουμε τη διευκόλυνση ε, συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe και να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση όσον αφορά την ε, θέση της Κομισιόν ότι δεν παίζει ο, ρο... τουρισμός κανένα ρόλο. Η Επιτροπή μας είναι υπεύθυνη και για τον τουρισμό και θα πρέπει να φροντίσουμε και στον τομέα αυτών που πάνε τα χρήματα και με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος, διότι είχαμε κάνει μια μελέτη και διαπιστώσαμε ότι, μόνο, ότι το 60% των ε, διαφθορτικών ταμείων πήγαιναν στους δρόμους και μόνο το 20% στους σιδηροδρόμους. Ε, θα πρέπει να προσέχουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα θα πρέπει να ε, πετύχουμε τους στόχους μας ε, και όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Ε, επειδή λοιπόν μιλάμε εδώ για πολλά χρήματα, πολύ ευχαριστώ, θα βάλω δύο-τρία επίθετα παραπάνω στο κείμενο, ώστε να είναι σαφές ποιοι είναι οι στόχοι μας και να μην αποτύχουμε όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Είδαμε μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ε, σε κάποιους τομείς, αλλά αύξηση σε κάποιους άλλους ε, και αυτό δεν είναι σκόπιμο. Επίσης, η μεταφορά είναι ξεχωριστό σημείο και μας ενδιαφέρει και ο τουρισμός είναι ξεχωριστό σημείο. Σας ευχαριστώ πάντως για την καλή συνεργασία και κατά τη διάρκεια της πέρασμένης εβδομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μάικλ. Ε, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Ωραία, έτσι ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε το χρόνο. Πέντε λεπτά διάλειμμα και κατόπιν θα συνεχίσουμε με τη συνεδρία των συντονιστών.